Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist äh, zwei Minuten nach neun. Είναι 9 και 2 η ώρα. Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε όλοι λάβει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Μία τροποποίηση υπάρχει. Το σημείο 8 θα συζητηθεί πριν το σημείο 5. Κατά τα άλλα δεν έχουμε επιθυμίες για τροποποίηση. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη και περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Έχουμε δύο έγγραφα με πρακτικά των συνεδριάσεων τη 27 η και 28 η Φεβρουαρίου και τη 20 η και 21 η Μαρτίου. Εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν έχουν ακουστεί αντιρρήσει, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Κατόπιν έχουμε το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Αποφάσεις των συντονιστών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες μας ε, κοινοποιούνται και σε εσά. Ε, και πάλι, εάν δεν ε, ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν οι αποφάσεις των συντονιστών. Και προχωράμε στο σημείο 4. Ως συνήθως, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Δηλαδή, από τη Λισαβόνα μέχρι το Ελσίνκι και από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρσοβία μας ακούνε. Και το Ανόβερο και το Λίνεμπουργκ ε, στην ε, κάτω Σαξονία και η Βαλένσια μας παρακολουθούν. Φροντίστε λοιπόν να αφαιρθείτε ανάλογα διότι όλα καταγράφονται. σχετικά με τις παρεμβάσεις σας. Ε, υπάρχει διερμηνία. Σας παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιες ανακοινώσεις. Η διάσκεψη στο Μαυρίκιο σχετικά με την διαφάνεια, η σύμβαση, συγγνώμη, ε, σύμφωνα με τη διαφάνεια στις διαδικασίες ISDS, ε, έχει τεθεί σε ισχύ. Έχει υπογραφεί από αρκετά κράτη-μέλη τώρα πια. Οι κανόνες UNCITRAL έχουν τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου. Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ. Ο 27ος γύρος των συστήσεων πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires. και το εμπορικό και το πολιτικό τμήμα συζητήθηκαν και στον επόμενο γύρο. Ο επόμενος γύρος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε μία ε, συνάντηση stock-taking ε, για να βολοσκοπήσουμε ε, την κατάσταση τον Μάιο. Επίσης, Ευρωπαϊκή Ένωση Νορβηγία, 5 Απριλίου στο Όσλο, θα συζητηθούν τα γεωργικά αγαθά. και μετά τη μετάφραση θα λάβει το έγγραφο, το σχετικό έγγραφο. Και επίσης ε, πραγματοποιήθηκε ο 18ος γύρος συζητήσεων ε, στο Τόκιο ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία στις 25 Απριλίου. Και εκεί συζητήθηκαν όλες οι πτυχές μιας εμπορικής σύμβασης στις δημόσιες συμβάσεις και τα γεωργικά αγαθά υπάρχουν ε, κάποια μικρά προβλήματα, διότι η Ιαπωνία έχει ξεκινήσει γεωργική μεταρρύθμιση και υπάρχει η ελπίδα να επιταχυνθούν οι εσωτερικές διαδικασίες ε, στη Ιαπωνία για να μπορέσουμε και εμείς ε, να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις μας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου και φτάνουμε τώρα στο νέο σημείο 5 στο παλαιό, το πρώην σημείο 8. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. Ε, πυρογνώμων μας είναι ο κύριος Ντάντι. Του δίνω κατευθείαν το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντάντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι ιδιαίτερα ε, ε, ειδικό, αλλά μου αρέσουν τα αλκοολούχα από τα Γι' αυτό ασχολήθηκα με το θέμα αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Η επισήμανση των προϊόντων σήμερα διασφαλίζει αξιόπιστη ενημέρωση και προσβάσιμη ενημέρωση για τους καταναλωτές. Βοηθά στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη στα προϊόντα. Σε εποχές ε, όπου οι αγορές είναι όλο και πιο συνδεδεμένες μεταξύ τους και αυξάνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επισήμανση. Να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντικέ είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις, ένα βασικό εργαλείο για την προστασία του διακριτικού χαρακτήρα και της ποιότητας των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύουμε ε, παραδοσιακές ε, γνώσεις ε, και τις σχετικές θέσεις εργασίας. Αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία υπεράσπιση ε, των ε, συμφερόντων στο πλαίσιο τη εμπορική πολιτικής στην Ευρώπη μέσω του οποίου προσπαθούμε ε, να παρέχουμε ανάλογη προστασία εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στι αγορέ των τρίτων χωρών για τα ευρωπαϊκά ποιοτικά προϊόντα. Η όλο και καλύτερη προστασία των προϊόντων με γεωγραφικέ ενδείξει πρέπει να συνοδεύεται από μια πιο αποτελεσματική στρατηγική προστασίας ε, και σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα στις τρίτες χώρες, ώστε να διαδικοποιηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης ε, της παραποίησης και της ε, δόλιας χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων. Επιπλέον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καταβάλουμε προσπάθειες για την όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας τους ή άλλου υπόψη τι ιδιαιτερότητε των διαφορών τομέων. γεγονό που θα μα βοηθήσει να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε πιο συνεκτική την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνε επίπεδο στον τομέα αυτών και ειδικότερα στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων ε, εμπορικών συμφωνιών με τρίτε χώρε. Α δούμε την πρόταση που συζητάμε σήμερα. Ο τομέα των αλκοολούχων ποτών είναι ένα από του σημαντικότερου ευρωπαϊκού τομεί ε, εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το 2016 αντιστοιχεί στο 8% των αγροδιατροφικών εξαγωγών της Ευρώπης μεταξύ των μεγάλων αγορών είναι η ΙΠΑ, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, ε, ο Καναδάς και η Κίνα. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ε, αξιοποίηση του τομέα. Βασικός ε, στόχος της πρότασης κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση της ισχύουσας νομοθεσίας με τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή μου όμως, η πρόταση κάνει κάποιες ε, ουσιώδεις τροποποίησεις που επηρεάζουν ε, τους τομείς αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής. Θα αναφερθώ σήμερα σε δύο πτυχές ειδικότερα. Πρώτη, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των ε, αλκοολούχων ποτών και δεύτερον ένα ηλεκτρονικό μητρό με όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά. Για το πρώτο σημείο θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει πάνω στι ετικέτε των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για εξαγωγή πέραν της γεωγραφικής ένδειξης ε, μία περαιτέρω μετάφραση που θα αναφέρει σε μια ε, ε, γλώσσα διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως προβλέπεται σήμερα τον ισχύοντα κανονισμό. Ο νέος κανονισμός θα προβλέπει αυτή τη δυνατότητα μόνο μέσω της υιοθέτηση από την Κομισιόν μιας κατεξοδότησης πράξης εφόσον ζητηθεί από την νομοθεσία μια τρίτη χώρα. Γεγονό που θα μπορούσε να έχει ω αποτέλεσμα μια πολύ αργή διαδικασία. Όσον αφορά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου, θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει ένα καινοτόμο και διαφανέ εργαλείο, αλλά κυρίω δυναμικό. Ταυτόχρονα, θεωρώ ότι η νομική του ισχύ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον κανονισμό. Το μητρό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιπλέον γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων τρίτων χωρών και προστατευόμενες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διεθνούς ε, συμφωνίας ε, σε περίπτωση που το επιθυμούν οι τρίτες χώρες αυτές. Θεωρώ ότι το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτε χώρε. Στο νου μου έχω τώρα χώρε όπω τι χώρε Μερκόσουρ που έχουν ήδη δώσει σημάδια ενδιαφέροντο προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και άλλε πτυχέ φυσικά, αλλά θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε ε, μετά από αυτήν εδώ την προκατακτική φάση. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις ε, των συναδέλφων και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω πρώτα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Κέλλη πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωθορίσω θερμά την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ασχολείται ακριβώς με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμεση των αλκοολούχων ποτών ε, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων. Νομίζω ότι η γενική δομή είναι κατάλληλη για τον τομέα αυτών και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει επιλεγεί συγκεκριμένη νομική βάση. Επίσης, το 95% της ε, παραγωγής ε, της Ιρλανδίας ε, καταλήγει σε 80 διαφορετικές αγορές και αντιπροσωπεύει μισό δισεκατομμύριο ευρώ που προστίθενται στην Ιρλανδική οικονομία κάθε χρόνο. Η εναρμόνιση των διαδικασιών για την καταχώρηση των αλκοολούχων ποτών και των γεωγραφικών ενδείξεων πηγαίνει ακόμα πιο πέρα και επικροτώ το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εισάγει τροποποιήσεις που θα επηρεάσουν την πρακτική, τις πρακτικές ε, κατά την παραγωγή. Κάποιες ε, στιλιστικές τροποποιήσεις ε, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Θα υποβάλω διάφορες τροποποίησεις για αυτές τις τροποποίησεις που στόχο έχουν να εξαλείψουν τις συγκρούσεις που υπάρχουν με την νέα διατύπωση και να διευκρινίσουν τις διατάξεις του νέου νόμου καθώς και τις σημαντικότερες δυσκολίες που δημιουργεί η νέα πρόταση. Ελπίζω οι συνάδελφοι να εξετάσουν με θετικό πνεύμα τις τροποποίησεις αυτές και ως Ιρλανδός χαίρομαι πολύ που συμμετέχω ε, στην εξέταση αυτού του θέματος. Η Φρεντερή Κερίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της που είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους επαγγελματίες που περιμένουν τα αποτελέσματα των δικών μας διαβουλεύσεων. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η πρόταση είναι ιδιαίτερα εκτενής και αναφέρεται και σε πολλά από τα σημεία εκείνα στο οποίο ήθελα και εγώ να αναφερθώ. Συμφωνούμε λοιπόν σε πολλά. Συνοψίζοντας για να μην επαναλάβω τα ίδια ε, προς ε, την Επιτροπή και τον εισηγητή μας. Είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω και η οποία έχει ακουστεί πολλές φορές και έχει να κάνει με τις εκτελεστικές ε, πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Σε ποιες κατηγορίες, ε, παράρτημα 3 για τις προστατευμένες ε, γεωγραφικές περιοχές, εδώ νομίζω ότι υπάρχει θέμα συζήτησης. Επίσης, δεύτερη παρατήρηση, η καταπολέμηση των αντιγραφών των προϊόντων μαϊμού είναι κάτι που πρέπει επίσης να κοιτάξουμε εδώ γιατί υπάρχει τέτοια παραποίηση προϊόντων, αλκοολούχων προϊόντων. Έχει αναφερθεί επίσης ξανά και ξανά η διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιούμε από το 2008 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για αλλαγές που μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τους παραγωγούς Μερικές φορές υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάλογα με τη χώρα. Κάποια αλκοολούχα ποτά, για παράδειγμα, που είναι από τη δικιά μου περιοχή, τη Βαλονία, που χρειάζονται έναν ορισμό αρκετά ελαστικό για να προστατευτούν και να προστατευτούν οι παραδόσεις που τα συνοδεύουν. Όλα αυτά σκοπεύω να τα συζητήσω με τον εισηγητή και θα υποβάλω και σχετικά τροπολογίες. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Να προωθήσουμε δηλαδή την τεχνογνωσία, να προστατεύσουμε την τοπική παράδοση, αλλά να διασφαλίσουμε και την προστασία των καταναλωτών που θέλουν να ξέρουν τι καταναλώνουν. Το οποίο, το λέω και εγώ, σε πολλά σημεία συμφωνούμε, αλλά προσοχή στις απομιμήσεις που μας έρχονται από διάφορες ασιατικές χώρες. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι αρμόδια επί της ουσίας για αυτό το θέμα. Συμμετέχω και εκεί ως ε, μέλος, οπότε και εκεί θα συνεχίσω τον αγώνα αυτό, κυρίως για την διατροφική αξία που είναι και αυτό ζωτική σημασία. Είναι κάτι που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό για τα αλκοολούχα ποτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα έπρεπε να προτείνει ήδη πριν από το 2014 έναν πίνακα σχετικά με αυτό. Αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πρόταση του Απριλίου του 2015 που ζητούσε ακριβώς με μεγάλη πλειοψηφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση για αυτά τα ζητήματα. Το αργότερο για το 2016. Είμαστε ήδη στο 2017. Η προ... πρότεινε 13 Μαρτίου να ε, μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά και να μεταφέρει τις προτάσεις της στους ε, επαγγελματίες. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί ένας τέτοιος κατάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές ε, δεν είναι ε, παρόντες. Χέλμουτ, ε, στο όνομα της κυρίας Φορένσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Φορένσα δεν είναι σε θέση να βρίσκεται εδώ σήμερα και γι' αυτό μου ζήτησε να σας μεταφέρω τις θέσεις της. Ως ΓΚΟΕ επικροτούμε την προσπάθεια να ε, εναρμονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με τα, τις, με τα νέα ε, μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τη νέα συνθήκη, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Και γι' αυτό προσπάθεια της ομάδας μας είναι να διατηρήσουμε το ισχύον επίπεδο προστασίας. Η βιομηχανία των αλκοολούχων ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας ε, και φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό που είπε η συνάδελφος μαζί με τις διαστάσεις, τις περιβαλλοντικές και τις επιπτώσεις στην υγεία. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, παραγωγή βιώσιμη και γι' αυτό χρειαζόμαστε σύγχρονη νομοθεσία που μπορεί να διασφαλίσει την προστιθέμενη αξία ε, και την απασχόληση στην Ευρώπη καθώς και να παρέχει στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αποφευθούν ε, οποιασδήποτε ενδείξεις μπορούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ε, και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της παραποίησης των προϊόντων. Δεν είναι εύκολο αυτό, γι' αυτό επικροτούμε διευκρινήσεις σε τομείς όπως είναι οι κανόνες που έχουν να κάνουν με τα συστατικά την ε, προαιρετική επισήμανση σχετικά με την ε, καταγωγή των πρώτων υλών κλπ. Θέλουμε να προωθήσουμε την ε, υπεύθυνη κατανάλωση και η σωστή επισήμανση είναι απαραίτητο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Επίσης, επικροτούμε την προσπάθεια να διευκρινιστούν οι κανόνες περί γεωγραφικών ενδείξεων. Και άκουσα ότι ο εισηγητής θέλει να επικεντρωθεί στο θέμα αυτό, θα συνεργαστούμε μαζί του στο θέμα αυτό. Το Μητρό Γεωγραφικών Ενδείξεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους μικρούς παραγωγούς και θα πρέπει να προωθείται η παραγωγή ε, και η πώληση των προϊόντων τους σε δίκαιη τιμή ώστε να μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Για το λόγο αυτό το Μητρό των Γεωγραφικών Ενδείξεων που ε, αντικαθιστά το παράρτημα 3 δεν θα πρέπει ε, να αποδυναμώσει την ε, διαφάνεια και τα πλεονεκτήματα του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα αφού εξετάσουμε και τις τροπολογίες. Ο συνήθως λέει πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ ο Ντέιβιτ. Um, ευχαριστώ πολύ. Ε, στον κύριο Κέλλη, ναι, εσείς φτιάχνετε το δεύτερο καλύτερο ουίσκι στον κόσμο μετά από αυτό που φτιάχνουμε εμείς, έτσι. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρότασή της και τον εισηγητή, τον κύριο Ντάντη, για την έκθεσή του. Τρία σημεία θέλω να θίξω, που έθιξαν κι άλλοι. Πρώτον, αυτό που είπε η κυρία Ρέις για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ε, κανόνες ε, για την ε, κατάσχεση τέτοιων απομιμήσεων. Αν μια εταιρεία υποψιάζεται πως έρχονται τέτοιες απομιμήσεις από την Ασία μέσω Ευρώπης για να πάνε στην Αφρική, δεν έχουν εντολή να κατάσχουν τα προϊόντα αυτά. Τώρα, για την ε, προέλευση και πώς αυτή καταχωρείται στις ετικέτες. Καταλαβαίνω ποια είναι η πρόταση, αλλά κατά τη γνώμη μου κινδυνεύουμε να δικηθούμε σε λάθος. Εγώ θα προτιμούσα την εθελοντική βάση που έχουμε μέχρι τώρα. Αν είναι blend το whisky, εντάξει, αυτό να υπάρχει. Αν πάρετε 5-6 τέτοια σκοτσέζικα, τα πάτε στη Γαλλία και γίνει εκεί... και γίνει εκεί η τότε η νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος για την μετάφραση, το είπε για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το είπε και ο εισηγητής. Φυσικά και χρειάζεται γεωγραφική ένδειξη πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν, αλλά ακριβώ εξαιτία των τοπικών ε, κανόνων και νομοθεσιών, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε υπόψη μας και τα τοπικά ονόματα. Δεν είναι θέμα το αν θα υπάρχουν ε, οι γεωγραφικές ενδείξεις, εντάξει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι τοπικές ονομασίες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να ενισχυθεί στην νομοθεσία. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι ένας κανονισμός που βοηθάει πολύ και θα συνεργαστώ με τον Νίκολα για να τον βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Ζωάν Φλόρ από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, Τμήματάρχης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ο τρέχον κανονισμός 110 έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλάδου. Τα αλκοολούχα ποτά είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γεωγραφικές ε, ενδείξεις επίσης γιατί ε, προσφέρουν ε, ακριβώς προστιθέμενη αξία στον κλάδο. Και είναι καλό λοιπόν να υπάρχει η κατάλληλη γεωγραφική νομική βάση. Ο κανονισμός αυτός είναι και ο τελευταίος στην κοινή γεωργική πολιτική προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν δεν σκοπεύει να αλλάξει οι κανόνες, απλώς να βελτιώσει τις νομοθετικές τάσεις και να φροντίσει να υπάρξει αυτή η ευθυγράμμιση. Τώρα, όσον αφορά τα όσα ανέφεραν οι ευρωβουλευτές για την πρόταση αυτή και για τη διαφορά ανάμεσα στη κατεξουσιοδότηση και τι εκτελεστικέ ε, πράξεις, εμείς ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε μια καλή ισορροπία και θα διατηρήσουμε ένα ελαστικό πλαίσιο. Πράγματι, χρειαζόμαστε ευελιξία. Από το 2009, 10 φορές Έχουμε τροποποιήσει τον κανονισμό 110, άρα αυτή είναι η απόδειξη ότι χρειάζεται ευελιξία. Και όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ε, γίνει επειδή τα κράτη-μέλη ζήτησαν να λύσουν κάποια πρακτικά ζητήματα τα οποία έπρεπε να λύσουν κατεπηγόντω. Όσον αφορά τις γεωγραφικέ ε, ενδείξεις, όντω ε, πρέπει αυτές να τι υπογραμμίσουμε και χρειαζόμαστε ένα πιο απλό σύστημα για να είμαστε στο ύψο των φιλοδοξιών μα. Έχουμε προβλέψει διατάξεις επίσης για τα πλαστά προϊόντα, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα. Το έχουμε κάνει και για τα αλκοολούχα ποτά. Όσον αφορά την καταγραφή, τις ακυρώσεις κλπ. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις διατάξεις όπως έχουν τώρα για τα αλκοολούχα ποτά. Ευχαριστούμε. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσει η Digitrade. Ναι, ευχαριστώ. Ε, ένα σύντομο σχόλιο. Η DG Trade ε, υποστηρίζει τον εξυγχρονισμό αυτών των διαδικαστικών πτυχών όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική, συνεκτική και διαφανή προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Εδώ έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό βήμα από πλευράς της DG Agri, το οποίο θα βοηθήσει ε, να προωθήσουμε το δικό μας σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο θέλουμε να αποτελέσει μοντέλο αναφοράς διεθνώς. Αυτές οι πιο αποτελεσματικές και διαφανείς ε, ε, διατάξεις ε, θα βοηθήσουν και στις διαπραγματεύσεις περί διατάξεων γεωγραφικών ενδείξεων στις Συμφωνίες Ελευθερών Συναλλαγών. Υποστηρίζουμε συνεπώς την πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σιγητά, κύριε Ντάντη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την σημαντική του συμμετοχή, τις ε, προτάσεις τους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ε, ενδιαφέρουσα δουλειά για το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας στις αρμόδιες επιτροπές. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Η κατεξοδότηση πράξη σίγουρα αποτελούν μια ευκαιρία πλούστευσης των διαδικασιών και αποφυγής ε, σχηνοτενών διαδικασιών όπως μας ε, υπενθυμίσατε πολλές φορές έχουν αλλάξει. Ε, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν τον τρόπο εργασίας μας και καταχώρησης αλλαγών ε, πιο απλό και για την είσοδο στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. Από αυτή την άποψη υποστηρίζουμε λοιπόν την ευκαιρία που μας δίδεται. Θεωρούμε ότι οι απλουστεύσεις πρέπει να είναι πραγματικές. Δεν μπορεί να γίνει όπως έγινε με την επισήμανση ε, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολο το να εξηγούμε σε μια άλλη χώρα ε, το τι περιλαμβάνει ένα προϊόν διατηρώντας ε, τη γεωγραφική ένδειξη στην αρχική γλώσσα. Όσον αφορά τις απομιμήσεις πρέπει να κάνουμε μια μάχη ε, χωρίς περιστροφές είναι θέματα που αφορούν εμάς στις αρμοδιότητές μας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς να υλοποιήσουμε μεθόδους που υπάρχουν και για άλλα αγροδιατροφικά προϊόντα που υποχρεώνουν τις χώρες ε, να αποσύρουν από τις αγορές αμέσως προϊόντα τα οποία είναι παραποιημένα. Ε, αυτό μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο κείμενό μας. Προς το παρόν σας ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις και συστάσεις σας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε μια σε βάθος έκθεση και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε εκτενώς το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η εξέταση του κειμένου θα γίνει 10-11 Ιουλίου μάλλον. Κλείνουμε έτσι το σημείο 5 της ημερησίας διάταξης και προχωράμε στο σημείο 6 που ήταν αρχικά το 5. Έχουμε την αποστολή στη Μάλτα στις 2 και 3 Μαρτίου. είχε προβλεφθεί αποστολή στη Μάλτα για να συζητήσουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά στο μεταξύ ε, μειώθηκε κατά ένα πρόσωπο η αποστολή εμένα. Μάλλον περιορίστηκε σε ένα άτομο η αποστολή σε μένα και είχαμε, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με το εμπορικό επιμελητήριο, να συζητήσω με ε, τα, το συνδικάτο, την ε, Συνομοσπονδία Εργατών, καθώς και να συζητήσω με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της, Μάλτα, της Μάλτας. Ε, ήταν παρούσα ολόκληρη η Επιτροπή, τέσσερα άτομα, και συζητήσαμε το θέμα των εμπορικών σχέσεων. Γενικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Μάλτα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο ο φόβος να αμφισβητηθεί ένα τέτοιο σύστημα, να διακυβευτεί λόγω του dumping από την Ασία ή ε, του προστατευτισμού στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, ο φόβος αυτός ήταν πολύ μεγάλος. Αναφέρθηκε ρητά η ανάγκη να έχουμε ένα εμπορικό σύστημα το οποίο να βασίζεται σε σαφείς κανόνες θα λάβετε αναλυτική έκθεση των ε, συνομιλιών. Σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Ε, αποστολή στην ε, Δυτική Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα. Το θέμα εδώ κυρίως ήταν οι εταίροι πώς βλέπουν την κατάσταση εντός της ΕΚΟΒΑΣ και πώς βλέπουν την ενδιάμεση EPA. Διαπιστώνουμε ότι και οι δύο χώρες όπου συνομιλήσαμε με τους ε, Υπουργούς Εμπορίου Οι δύο χώρες λοιπόν αυτές ε, θεωρούν ότι η νέα συμφωνία είναι χειρότερη από αυτήν της ΕΚΟΒΑΣ και οι δύο χώρες αυτές όμως θέλουν να διατηρήσουν την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γι' αυτό ε, υπέγραψαν. Και αυτή η θέση διέπει όλες τις συζητήσεις και στα think tanks και ε, στις ε, νομοσπονδίες εργατών. Τη θέση αυτή λοιπόν ότι αυτή η καινούρια EPA είναι χειρότερη από την προηγούμενη, την υπογράψαμε όμως γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε την πρόσβαση στην αγορά, αυτή η θέση ε, υπήρχε γενικά παντού. Και λόγω της σταθεροποίησης στην περιφέρεια αυτή, νέα κυβέρνηση στην Κάνα, σχετικά νέα κυβέρνηση στην Ακτή Ελεφαντοστού, νέα κυβέρνηση στην Κάμπια, ε, στη Μαυριτανία. Σύντομα θα υπογραφεί λοιπόν ε, αυτή η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και ελπίζουμε και η Νιγηρία να υπογράψει. Η οποία ε, αντιμετωπίζει προβλήματα επειδή η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση υψηλού επίπεδου και οι δύο χώρες ελπίζουν να ολοκληρώσουν σύντομα την ε, διαδικασία της ε, Συμφωνίας Εταιρικής ε, Σχέσης ΕΚΟΒΑΣ, μέχρι το 2020 δηλαδή, διότι τότε θα τεθούν σε ισχύ οι εξωτερικοί δασμοί, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά τις Προσωρινέ ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης. Από εκεί και πέρα ε, τίθεται και το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και γενικά Όσον αφορά την παραγωγή της μπανάνες δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Στον ε, ανεπίσημο τομέα όμως, στο ανεπίσημο τμήμα, την ε, παραγωγή κακάο για παράδειγμα, οι συνθήκες εργασίας ε, είναι πολύ κακές. Και ελπίζουμε οι συνθήκες να βελτιωθούν με τη συνεργασία μας ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση σχετικά με τους κανόνες FLECT στην Γκάνα. Στο μεταξύ η Ινδονησία έχει προσπεράσει την Γκάνα στο θέμα αυτό. Η διαφορά όμως είναι ότι η Γκάνα την βιώσιμη δασοκομεία ε, την θέλει όχι μόνο για το εξωτερικό εμπόριο, αλλά και για την ε, Γκάνα αυτή καθ' αυτή. Είναι λοιπόν πολύ θετικό το ότι προωθείται έτσι η βιώσιμη δασοκομεία γενικά. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν επιτυχημένη αυτή η αποστολή. Ιδιαίτερα συνομιλήσαμε με τον Υπουργό Εμπορίου της Γκάνα που είναι εμπειρογνώμων στο θέμα αυτό. Ως ε, γενικός γραμματέας ε, του ΠΟΕ γνωρίζει ιδιαίτερα καλά τα θέματα αυτά και παρακολουθήσει τη συνέχεια της διαδικασίας για να καταλήξουμε σε συμφωνία εταιρικής Πάντως απομένει δουλειά να γίνει. Αυτά από μένα. Ε, διάφοροι συνάδελφοι ε, ασχολήθηκαν επίσης με το θέμα που θέλουν κάτι να προσθέσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θέλω να πω εδώ ότι η επίσκεψη αυτή, αυτό το ταξίδι δηλαδή, ήταν πολύ ενδιαφέρον και μάθαμε πάρα πολλά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αξία της αποστολής αυτής, αυτού του ταξιδιού, ήταν, όπως πάντα, ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με πολλούς εταίρους. Δεν συναντάμε δηλαδή μόνο τους πολιτικούς, δεν πάμε να δούμε μόνο τους βουλευτές ή τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά ε, στην πραγματικότητα όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, έχουμε συναντήσεις με εκπροσώπους από διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Από την κοινωνία των πολιτών συναντιόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και συναντάμε επίσης και εκπροσώπους των συνδικάτων βλέπουμε και εκπροσώπους των εργοδοτών επίσης. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την άποψη όλων και όχι μόνο μερικών έτσι επιλεγμένα. Και βέβαια οι απόψεις που ακούμε είναι διαφορετικές μεταξύ τους πολύ συχνά, αποκλίνουν. Συνεπώς έχουμε ένα ολόκληρο εύρος απόψεων και στη συνέχεια είναι πιο εύκολο έτσι να καταλήξουμε και εμείς σε κάποια συμπεράσματα. Όμως τα συμπεράσματα από το ταξίδι αυτό είναι τα εξή, κατά τη γνώμη μου. Στις περισσότερες συνομιλίες που είχαμε, ακούσαμε ότι οι σταθερές συμφωνίες είναι προτεραιότητα από προσωρινές τοπικές συμφωνίες. Αλλά οι εταίροι μας είναι πολύ ευχαριστημένοι που έχουν τη δυνατότητα να έχουν τέτοιες προσωρινές συμφωνίες. Και γιατί, γιατί χωρίς αυτές τις προσωρινές συμφωνίες η κατάσταση των χωρών αυτών θα ήταν ακόμα χειρότερη. Και σας υπενθυμίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χώρες με έναν προϋπολογισμό ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτάται από μία μόνο κατηγορία εσόδων. Έσοδα δηλαδή που προέρχονται από εξαγωγές πρώτων ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Οπότε κάθε αστάθεια, κάθε αλλαγή, ακόμα και πιο μικρή, κάθε δυσκολία εξαγωγών που προέρχεται από τη δικιά μας την πλευρά, για αυτές τις χώρες σημαίνει ένα πραγματικό κίνδυνο, σημαίνει πολύ καταστροφικές συνέπειες πολύ βαριές για αυτούς. Τέτοιες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις στη συνέχεια καταλήγουν σε κοινωνικό χάος τους δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι πάντα υπέρ τέτοιων προσωρινών συμφωνιών και χαίρομαι που το ίδιο πιστεύουν και οι εταίροι μας εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, που συζητήσαμε και επί τόπου. Θα έπρεπε εδώ να καθίσουμε και να σκεφτούμε και να συζητήσουμε κατά πόσο οι περιφερειακές συμφωνίες εξακολουθούν να έχουν νόημα ή εν πάση περιπτώσει αν πρέπει πάντα να στοχεύουμε σε τέτοιες συμφωνίες. Και θέλω εδώ να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Για χρόνια και χρόνια διαπραγματευόμαστε και μετά καταλήγουμε σε συμφωνίες οι οποίες δεν ισχύουν γιατί μια ή δύο χώρες δεν θέλουν να τις ε, προσυπογράψουν Οπότε τελικά έχουμε χάσει τόσο χρόνο, έχουμε ζητήσει τόσα πράγματα, χωρίς όμως τίποτα να υλοποιείται τελικά. Και γιατί, γιατί είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Όλες αυτές οι χώρες, πρέπει να το πούμε, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έχουν διαφορετικές παραδόσεις, ιστορία, θρησκεία, επίπεδο ανάπτυξης, μέγεθος κλπ. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Νιγηρία εκείνη η οποία θέλει πιο πολύ να προχωρήσει και είναι μια χώρα που θεωρεί ότι μπορεί να έχει πολλές προοπτικές και ότι είναι μια ισχυρή χώρα. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο σε βάθος. Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο χωρών που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους όπως σας είπα μέσα στις οποίες υπάρχουν κάποιες που θέλουν τις περιφερειακές συμφωνίες, άλλες δεν τις θέλουν ή κολλησιεργούν, ε, τελικά τι πρέπει να κάνουμε. Μήπως θα έπρεπε βασισμένοι στις εμπειρίες μας να πάμε να μιλήσουμε και με αυτούς που δεν θέλουν. Γιατί ίσως θα καταφέρουμε να τις πείσουμε ότι τελικά είναι και προς δικό τους όφελος τέτοιες συμφωνίες. Να μιλήσουμε λοιπόν και με αυτούς που τις απορρίπτουν. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουτ Σόλ. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Όσον αφορά αυτήν την τελευταία πτυχή που ανέφερε ο συνάδελφο Σίνφελτ, είναι πολύ ενδιαφέρον το, το θέμα αυτό. Και συμφωνώ και με σένα και με εκείνον ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη. Πολλά μάθαμε. Αλλά έτσι φτάνουμε και στο ερώτημα η συνολική οικονομική ικανότητα πώς επηρεάζει τις σχέσεις με τους εταίρους μας. Και εμείς είμαστε μία κοινότητα που ε, προβάλλει το κοινό συμφέρον απέναντι στους εταίρους μας. Είμαστε λοιπόν μία μονολυθική ένωση, ένας μονόλυθος ή καταφέρνουμε να, ε, να συνδυάσουμε τις διάφορες θέσεις και τα διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν και τι επιπτώσεις έχει αυτό προς τα έξω. Οι χώρες ε, της Αφρικής, λοιπόν, ε, τι θέση έχουν απέναντι στον ΠΟΕ και τι δυνατότητες έχουν για περιφερειακή συνεργασία γνωρίζοντας τις συχνά πολύ αντιφατικές προϋποθέσεις που υπάρχουν εντός των διαφόρων χωρών. Και ας πάρουμε για παράδειγμα την Νιγηρία. Και ε, στην περιφέρεια αυτή της Αφρικής ε, υπάρχει σημαντικό χάσμα ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Και είχαμε τη συζήτηση εδώ για τους κανόνες FLECT. 30.000 άνθρωποι στις γειτονικέ χώρες, ε, στο Μάλι, στην Μπουρκίνα Φάσο και λοιπά. Ε, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να έχουν εισόδημα από την δασοκομεία ή με νέες φυτίες μπανάνας ή κακάο. Και αυτή είναι μια διαδικασία με την οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις καταστάσεις αυτές και στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Δύο παρατηρήσεις ε, λοιπόν ε, σχετικά με τις ε, συνομιλίες. Στην συζήτηση που είχαμε στο Κοινοβούλιο στην ακτή Ελεφαντοστού, διαπιστώσαμε ότι οι βουλευτές εκεί δεν ήταν τόσο καλά ενημερωμένοι όσο είναι απαραίτητο για κάποιον που έχει τη θέση αυτή. Το θέμα λοιπόν της διαφάνειας της ενημέρωσης ε, των βουλευτών από πλευράς της κυβέρνησης είναι απολύτως απαραίτητη. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πίεση ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Και η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ο διεθνής ανταγωνισμός έχει άμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς στην περιοχή αυτή. Για παράδειγμα, στην παραγωγή μπανάνας. Είναι σαφές ότι η περαιτέρω μείωση της τιμής της μπανάνας θα καταστήσει μη επικερδή την παραγωγή και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση ε, παράδοξη. Η παραγωγή λοιπόν ε, των ε, Ευρωπαίων παραγωγών έχει επιπτώσεις και στην παραγωγή της Αφρικής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε τη διαμόρφωση τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια. Θέλουμε να προωθήσουμε την απασχόληση και θα πρέπει ε, την κοινοβουλευτική συνέλεση του ΠΟΕ να την εκμεταλλευτούμε για να συζητήσουμε με τους συναδέρφους τα θέματα αυτά. Ήταν ε, λοιπόν ε, πολύ χρήσιμη επίσκεψη αυτή και λυπάμαι που δεν ήταν μαζί μας ο εισηγητής. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη. Πολλά σημείωσα, αλλά νομίζω ότι το κύριο μάθημα ε, για την ΕΚΟΒΑΣ ε, έχει να κάνει με την Ιγυρία που είναι τόσο σημαντικός παράγοντας στην περιοχή αυτή έτσι ώστε εάν η Νιγηρία δεν θέλει να συμμετέχει ε, σε ε, συμφωνία εταιρική σχέσης ε, ή ελεύθερο εμπορίου με την, στο πλαίσιο της ΕΚΟΒΑΣ, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης έχει βελτιωθεί πολύ από την αρχική εκδοχή που είχαμε. Ε, κάτι που σχετίζεται με τις συζητήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 50 είναι το θέμα των ποσοστώσεων ε, και ιδιαίτερα όσον αφορά την μπανάνα. Στον ΠΟΕ είχαμε 15 ετή εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, την Νότια Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το όλο θέμα των δασμολογικών ποσοστώσεων είναι πολύ ευαίσθητο. Αυτό σχετίζεται πολύ με τις συζητήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 50, διότι νομίζω ότι ε, η Μεγάλη Βρετανία ε, απορροφάει το 44% της συνολικής ποσόστοσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν αποχωρήσει η Βρετανία θα πάρει μαζί της την, την ποσόστοση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ίδια ποσόστοση. Ε, θα ήταν πιο γενναιόδωρο να έχει το Ηνωμένο Βασίλειο δική του ποσόστοση. Αλλά αναφέρθηκαν αρκετές φορές οι ποσοστώσεις ε, και νομίζω ότι το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει, θα το θίξουν οι χώρες αυτές. Σε διάφορες αποστολές ε, έχω συζητήσει το θέμα αυτό και πάντα αναφέρονταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις. Η κατανομή λοιπόν των ποσοστώσεων αυτών, όπως για παράδειγμα το αρνί της Νέας Ζηλανδίας, ε, από το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο απορροφά το 50%, νομίζω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό θέμα στις διαπραγματεύσεις. Και όπως ε, είπε και ο πρόεδρος, ε, έχουμε την συμφωνία ΣΥΤΑ. Εγώ θα ήμουν υπέρ μιας τέτοιας υπερσυμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά. Όλα αυτά τα θέματα πάντως εθίχτηκαν πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται η παραγωγή κακάο και μπανάνας καθώς και η συνάντηση με τον ε, Υπουργό Εμπορίου καθώς και με τους βουλευτές ε, ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι η επίσκεψη αυτή επικεντρώθηκε σε πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις ε, που να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Και τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στην οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι ήταν σημαντική αυτή η αποστολή. Θα λάβετε την αναλυτική έκθεση. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω στο θέμα αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά τις μελλοντικέ συμφωνίες. Και αναφέρθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Ωραία, κλείνω το θέμα αυτό και φτάνουμε τώρα στο σημείο 8, το αρχικό 7 δηλαδή, που επίσης σχετίζεται κάπως με την αποστολή αυτή. Ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ και στην ακτή Ελεφαντοστού και στην Κάνα ήταν η διαφθορά και κατά την ε, κατανομή γης ε, και, κατά, ε, και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο που θα το συζητήσουμε αυτό. Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε, τρεις, σε τρίτες χώρες και η συντάκτρια της νομοδότησης είναι η Καρολίνε Κρασφάντερ. Ευχαριστώ Μπέρντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ταιριάζει πολύ καλά το θέμα αυτό στην ε, συνολική μας συζήτηση. Ακούσαμε ότι υπάρχει διαφθορά σε πολλούς τομείς. Είναι κάτι που επηρεάζει ε, αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οδηγεί σε ανισότητα. Διακυβεύεται έτσι η κοινωνική δικαιοσύνη και έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Στην γνωμοδότησή μου επικεντρώθηκα στα εξής θέματα. Ε, την ε, δέσμευση με διεθνείς ε, συμβάσεις κατά της διαφθοράς, να υπάρχουν ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες, η ενεργό συμμετοχή μη κυβερνητικών παραγόντων και νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικές πτυχές επιπλέον. Λείπουν οι μηχανισμοί για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι διατάξεις ε, κατά της ε, διαφθοράς ε, και για να μπορέσει να υπάρξει εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε δεσμευτικά μέτρα, διότι η εθελοντική προσέγγιση δεν θα μας βοηθήσει αρκετά και γι' αυτό στην γνωμοδότηση λέω σαφώς ότι σε μελλοντικές συμφωνίες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ρήτρε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι εμπορικοί μας εταίροι δεν τηρούν αυτές τις διατάξεις, θα πρέπει να αναστέλλεται η εμπορική συμφωνία ή να επιβάλλονται κυρώσεις. Δεν είχα πολύ χρόνο, δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω όλες τις ε, σημαντικές πτυχές, ε, γι' αυτό θα υποβάλω και κάποιες ε, τροπολογίες. Στις τροπολογίες με ενδιαφέρει η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η επιβολή των μέτρων κατά της διαφθοράς, αλλά να υπάρχει και διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες. Επιπλέον, θεωρώ σημαντικό να υπάρχει ανεξάρτητος ε, φορέας παρακολούθησης. Η άφετη είναι αρμόδια επί της ουσίας και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν χθες. Ε, υπέβαλα λοιπόν έχω κάποιες τροπολογίες οι οποίε όμω επικαλύπτονται εν μέρη με το περιεχόμενο τη νομοδοτησή μου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τι προτάσει των συναδέλφων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζάχη από το ΕΛΚ, η Σκιώδη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Συγητρία για το σχέδιο έκθεσης. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι σημαντικότατο θέμα και επιτέλους ε, πρέπει να ενταχθεί και στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δουλειά που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της TTIP η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα. Καλό θα ήταν στο εξή να διαπραγματεύεται διατάξεις καταπολέμησης διαφθοράς η Κομισιόν σε όλες τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Έχει γίνει αυτό ήδη στη συμφωνία με το Μεξικό και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Επιβεβαιώνεται, όπω έχετε αναφέρει στη στρατηγική εμπόριο για όλου, ότι διατάξει τέτοιε θα συζητούνται και στις μελλοντικέ νέες διαπραγματεύσεις. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη-μέλη πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς στις διαπραγματευτικές εντολέ που αναθέτουν στην Κομισιόν. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεση. παρουσιάστηκε από την εισηγήτρια, την ευχαριστούμε και θα υποβάλουμε συμπληρωματικές και διευκρινιστικές τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε στο ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην πρόθεση της χρηστής διακυβέρνησης και των αξιών μας. Θέλουμε επίσης να διευκρινίσουμε πόσο σημαντική είναι η συνοχή μεταξύ των εμπορικών πολιτικών της Ένωσης και του κοινοτικού κεκτημένου, κυρίως σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό θα, το κεκτημένο θα πρέπει να αποτελεί βάση αναφοράς στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, συμμεριζόμαστε την ιδέα που δίνει το κείμενο ε, για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στο θέμα αυτό. Σε γενικότερο επίπεδο πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ενισχύσει την ε, διεθνή συνεργασία και να αποτελέσει πρότυπο ηγεσία στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Μην ξεχάσουμε ότι το SPG ΣΥΝ απαιτεί υπογραφή και επικύρωση τη ε, Σύμβαση των ΗΕ για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε επακριβώ ε, την υλοποίηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το ECR ο κύριος Κάμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς αναγνωρίζουμε στο ΙΣΙΑΡ ε, πόσο αρνητικά επηρεάζει το εμπόριο η διαφθορά. Αποθαρρύνει τις επενδύσεις, προωθεί την του ανταγωνισμό και στρεβλώνει τις ε, ε, δημόσιες συμβάσεις και τις σχετικέ διαδικασίες. Η διαφθορά κατά την άποψή μου τίνει να συμβαδίζει με τα, δημογραφικά, με τα συγγνώμη, γραφειοκρατικά προσκόμματα πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προβλήματο αυτού και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται διατάξει αντιμετώπιση τη διαφθορά σε μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε. Πρέπει να αποτελεί προέχον θέμα, προεξέχον θέμα σε μελλοντικέ ε, διαπραγματεύσει, ε, να συνάδουν με τι εξωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και με τη στρατηγική εμπόριο για όλου. Ε, καλωσορίζουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών του ιδιωτικού τομέα και λοιπόν ενδιαφερομένων στην υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης διαφθοράς και των σχετικών διατάξεων σε εμπορικές συμφωνίες. Ε, υποστηρίζουμε τη δημιουργία λοιπόν εργαλείων που θα παρέχουν καλύτερη κατεύθυνση και θα προωθούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Καλωσορίζουμε τις ε, απόψεις της εισηγήτρες και θέλουμε να προσθεθούν και περαιτέρω συστάσεις κατά πολέμησης διαφθοράς μέσω του εμπορίου όπως ε, διαδικασίες ε, αντιμετώπισης ε, των και εξέταση ανείχνευση των χρηματοοικονομικών ροών. Θέλουμε ωστόσο να επισημάνουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις διότι η διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν συνεπάρχουν πάντα. Ορισμένε πρακτικέ διαφθορά δεν έχουν απαραίτητα επιπτώσει στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω συμβαίνει σε περιπτώσει διαφθορά μεταξύ ιδιωτών. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυσικά οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά στι εμπορικέ ε, συμφωνίε, αλλά δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπορικό εμπόδιο. Εδώ μιλάμε για εμπόριο και όχι για πολιτικές, οπότε πρέπει να κεντρωθούμε στη διευκόλυνση του εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι στην αίθουσα. Θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφος μου Δίτα που ήταν ε, ε, Σκιώδης δεν, είναι, δεν ήταν εδώ σήμερα, θα σας διαβάσω τις απόψεις της. Χαιρέτε που η συγγήτρια επισημαίνει ότι η σύνδεση μεταξύ διαφθορά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η καταπολέμηση τη διαφθορά θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό φυσικά περιλαμβάνει τον τρόπο ε, που θεωρούμε ε, του κανόνε του διεθνού εμπορίου. Εμείς ε, συμφωνούμε με το περιεχόμενο της εκθέσης, αλλά θέλουμε να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ διαφθοράς και επιχειρηματικού περιβάλλοντος ε, και να αναφέρονται και τα βήματα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφθορά είναι σημαντικό πρόβλημα για την οικονομία και την κοινωνία μιας χώρας. Δυσκεραίνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όχι μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους εγχώριους επιχειρηματίες. Επειδή η διαφθορά εμφανίζεται και στα τελωνία, ε, στους κανονισμούς αδειοδότησης ε, επηρεάζει σημαντικά τις εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες των ε, ευρωπαϊκών εταιριών και σε τρίτες χώρες. Η διαφθόρα φυσικά εμποδίζει την μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο των GSP και των σχετικών συμφωνιών ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τη διαφθόρα και είναι σημαντικό να ληφθούν σημαντικά βήματα στο πλαίσιο των διαφόρων συμφωνιών. Ε, Δεδομένη τη αναθεώρηση του GSP που πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι μια ευκαιρία. Οι εμπορικέ συμφωνίε μπορούν μεν να ορίσουν πρότυπα τη διαφάνεια, ε, αλλά δεν είναι τα μόνα εργαλεία. Υπάρχουν και πιο πολιτικά εργαλεία και συμφωνίε όπω η Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία ή οι Συμφωνίες ε, Σύνδεσης και αυτά τα ε, εργαλεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που λένε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι παρά ένας κρίκος μιας ε, μεγαλύτερης αλυσίδας. Οπότε θα, κάνουμε, θα υποβάλουμε τις σχετικές τροπολογίες ε, για το κείμενο. Ευχαριστούμε Μαρίτια. Helmut Ευχαριστώ. Θέλω να μεταφέρω το μήνυμα της δικιάς μας κοιόδου συζητήριας που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Υπογραμμίζει και λέει προς την ε, συντάκτα της γνωμοδότησης ότι χαιρόμαστε για αυτήν την γνωμοδότηση που συνδέει τη διαφθορά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. που συνδέεται τη διαφθορά με παραβιάσεις περιβαλλοντικού τύπου, ποιότητα ζωής κλπ. Και θέλει να υπογραμμίσει ότι αυτά τα τελευταία πολύ συχνά χρησιμοποιούνται οι εμπορικές συμφωνίες ανάλογα με το πώς διατυπώνονται και αν δεν έχουν ε, ρήτρε κατά της διαφθοράς που όμως δελοποιούνται και όλα, τότε αφήνουν τη διαφθορά να ανθίσει. Αυτή είναι η άποψη που θέλουμε να μεταφέρουμε στην Επιτροπή μας. Επίσης, η νομοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες παράνομες ε, τέτοιες δραστηριότητε θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε για εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. δεν θα πρέπει να αφήνουμε κανένα παράθυρο ανοιχτό για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Και συμφωνώ με τους συναδέρφους που υπογραμμίζουν το θέμα της διαφάνειας, των κανόνων για διαφάνεια, δηλαδή που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες, ότι είναι στοιχείο κλειδί. Τώρα για την μακροοικονομική αρρωγή προσθέτω ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι σε κάθε εμπορική συμφωνία. Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ και θα συνεργαστούμε με την συντάκτρια της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριος γιαντλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω κύριος Σένφελτ. Εδώ συζητούμε για μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Πολύ σωστά ο Πρόεδρος είπε ότι συνδέεται με το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε. Εκείνο δηλαδή που έχει να κάνει με την επίσκεψή μας στην ακτή Λιφαντοστού και την Κάνα. Η διαφθορά αποτελεί πολιτική μάστιγα και κοινωνική μάστιγα. Είναι κάτι σαν μια αρρώστια που έχει καταστροφικές συνέπειες και εμποδίζει τις χώρες να αναπτυχθούν. Κυρίως τις πιο φτωχές ακριβώς χώρες και τις λιγότερο αναπτυγμένες. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να βγούνε. Αλλά είναι και κάτι πολύ σημαντικό για μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Διότι είμαστε από τους μεγαλύτερους δωρητές στον κόσμο είμαστε από αυτούς που δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουμε τις υποανάπτυξη χώρες και τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Αναφερθήκαμε στις εμπορικές συμφωνίες, στις επενδυτικές συμφωνίες, σε όλες τις οικονομικές πτυχές. Ναι, πράγματι πιστεύω ότι ακριβώς εκεί είναι και το πιο σημαντικό εργαλείο που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε ε, τις χώρες. Η άμεση οικονομική αρρωγή επίσης υπάρχει. Στην Αφρική, για παράδειγμα, εμείς δίνουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην Αφρικανική Ήπειρο. Δυστυχώς, ένα κομμάτι των χρωμάτων αυτών δεν πηγαίνει στους δικαιούχους, εκεί που πραγματικά απευθύνεται, και ακόμα και αν φτάσει στον προορισμό του το χρήμα αυτό, δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ένα ζήτημα τεράστια σημασία. Είναι λοιπόν προ το συμφέρον της Ευρωπαϊκή Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει τεράστια ποσά, είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε πώ χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα, να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμω είναι και προ το συμφέρον των ε, χωρών αυτών τις οποίες βοηθούμε και έχουμε μαζί τους πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Γιατί οι χώρες αυτές πρέπει να αποτελούν αξιόπιστο εταίρο για μας. Και άρα να ξέρουμε ότι καταπολεμούν τη διαφθορά, τη μειώνουν. Ό,τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι πραγματικά αναγκαία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ορίζουμε το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Όντως, μας δίνει τροφή για σκέψη για το δικό μας το έργο και για το πόσο θα προχωρήσουμε σε περισσότερες διατάξεις κατά της διαφθοράς. Όπως ανέφεραν ήδη πολλοί ευρωβουλευτές, Εννοείται ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την καταπολέμηση του φαινομένου και το έχει πει και τον Οκτώβριο του 2015 στην ανακοίνωσή της ξανά και ξανά μάλιστα από τότε. Ήταν τότε που ξεκινήσαν διαπραγματεύσεις για το TTIP, αλλά όπως λέμε στην ανακοίνωσή μας η ιδέα ήταν να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες. Και όπως είπε και η κυρία Σαϊφή, αν σκοπεύει να τα συμπεριλάβει σε μελλοντικέ συμφωνίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, και το έχει ήδη κάνει με τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με το Μεξικό, για παράδειγμα. Θέλω να διευκρινίσω δηλαδή ότι πράγματι αυτό που κάνουμε και εμείς είναι να προτείνουμε κάτι τέτοιο στις μελλοντικέ συμφωνίες. Επίσης, χαιρόμαστε και από προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Λάγκε και της Επιτροπής αυτής, ήδη από πέρυσι, και είναι πράγματα τα οποία ελοπίθηκαν και γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του Μεξικό. Όπως αναφέρει το σχέδιο γνωμοδότησης και η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, είναι κάτι που συνδέει τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη διαφθορά. Η σχέση αυτή είναι πράγματι ζωτική σημασίας. Και παλιότερα έχουμε διαπιστώσει ότι η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου και την χρηστή διακυβέρνηση και σίγουρα είναι ένα τεράστιο βάρος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως είπαν πολλοί ευρωβουλευτές ήδη, πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες και γι' αυτό και θέλουμε και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι φυσικά και υπάρχουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες στα πλαίσια της συμφωνίας GSP-SYN και όπως ξέρετε η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για την ε, επικύρωση και την υλοποίηση διαφόρων διεθνών συμβάσεων μεταξύ άλλων και των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Από το 2014 και μετά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν ε, εκπονήσει ένα σχέδιο, έναν μηχανισμό καλύτερα ελέγχου της υλοποίησης της συμφωνίας αυτής με γραπτές ερωτήσεις, με κάτι σαν βαθμολόγιο και βέβαια και με επισκέψεις επιτόπου. Η δεύτερη έκθεση για την συμφωνία αυτή, που αναφέρεται και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα τέλη της χρονιάς αυτής, από όσο γνωρίζω. Και όπως επίσης έχει ήδη υποθεί, κάνουμε την σύνδεση αυτή ήδη ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την διαφθορά στη Συμφωνία του Κατονού. Εκεί το άρθρο 9 αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχέση τους με την διαφθορά. Και υπάρχει και σχετική διαδικασία στο άρθρο 97 της Συμφωνίας Κοτονού για να αρχίζουν διαβολεύσεις άπαξ και εντοπίζονται περιπτώσεις διαφθοράς. Όσον αφορά τώρα το έργο μας για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και πώς συμπεριλαμβάνουμε το θέμα της διαφθοράς σε αυτές, εδώ όπως ανέφεραν και κάποιοι ευρωβουλευτές ήδη, θέλω και εγώ να πω ότι οι εμπορικές συμφωνίες διέπουν εμπορικές σχέσεις, οπότε το οικονομικό σκέλος σε σχέση με τη διαφθορά μπορεί να υπογραμμιστεί. Είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο δυσκολεύει, εμποδίζει το εμπόριο και εμποδίζει την ισότιμη σχέση και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμω, συγχρόνως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στις εμπορικές συμφωνίες φυσικά και πρέπει να ε, ασχολούμαστε με το θέμα της διαφθοράς σε εμπορικές συμφωνίες και υπάρχουν καλά παραδείγματα, για παράδειγμα στις δημόσιες συμβάσει, στα τελωνία, όπως επίση ανέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτέ ήδη. Και εκεί φροντίζουμε και εμεί να συμπεριλάβουμε το θέμα τη διαφθοράς. Τώρα, την βασική γραμμή της προσέγγισής μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς ανάμεσα τους εσωτερικούς κανόνες, το κεκτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι κάνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η βασική μας κατευθυντήρια γραμμή είναι η σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, που έχει επικυρωθεί ήδη από όλε τις χώρες μέλη, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια. Όταν κοιτάμε όμως τις διάφορες διατάξεις και τις προδιαγραφές, πρέπει να δούμε και κατά πόσο έχουμε ήδη αρκετές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ευρωπαϊκό ε, κεκτημένο που να μπορούμε να υποστηρίξουμε στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία των καταγγελόντων, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Και ξέρω ότι έχει ασχοληθεί με αυτό ε, συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δούμε προσεκτικά πώς θα προωθήσουμε εμπορικές συμφωνίες. Όπως ξέρετε δεν υπάρχουν ακόμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινά αποδεικτοί κανόνες για την προστασία των κατεγγελόντων. Έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις, γίνεται δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταλήξουμε σε πρόταση και περισσότερες ιδέες από αυτού μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Αυτό όμως συγχρόνω σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με κάτι τέτοιο όταν πρόκειται για εμπορικέ συμφωνίες. Όσον αφορά τώρα την επιβολή, τη συμμόρφωση, δηλαδή και την απώλεια κερδών. Εδώ θέλω να πω ότι αν δείτε την συμφωνία GSP, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και μονομέροι μέσα. Υπάρχουν, ε, υπάρχει θέμα ισορροπίας εδώ και πρέπει να δούμε πώς ε, το θέμα της ε, συμμόρφωσης θα το δούμε σε σχέση με το τι ισχύει στο ποινικό δίκαιο. Σκοπεύουμε σύντομα να έρθουμε με πιο συγκεκριμένες προτάσεις τους επόμενους μήνες και προσβλέπουμε σε ανταλλαγή απόψεων σε βάθος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι ετοιμάζονται και εργαστήρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και το εμπόριο. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για μας προκειμένου να διατυπώσουμε την προσέγγισή μας. Προσβλέπουμε στις επόμενες συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστούμε. Καρολίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές ε, προτάσεις που ακούστηκαν. Στόχος είναι να έχουμε αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς ε, εντός της Ευρώπης ε, σε σχέση με τρίτες χώρες. Μάλλον σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις τρίτες χώρες και Γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα να έχουμε υποχρεωτικούς κανόνες, διότι αλλιώς δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Επίσης πρέπει να έχουμε σωστή επιτήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ε, αυτών των ε, μέτρων ε, και είναι σημαντικές για μένα και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικό και το θέμα της προστασίας των κατακελώντων, κάτι που θα πρέπει να ρυθμιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να το ζητήσουμε και στις εμπορικές συμφωνίες. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία και περιμένω να δω και τις ε, πολλέ και ενδιαφέρουσε τροπολογίες σα και θα προσπαθήσω όλες να τις ε, υιοθετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. 8 Μαΐου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στις 13 Μαΐου. Φτάνουμε στα σημεία 9 και 10. Κοινή συζήτηση σχετικά με την συμφωνία με την Κούβα. Γνωμοδότηση για ε, την ΑΦΕΤ και δίνω κατευθείαν το λόγο στον ε, εισηγητή τον κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη συζήτηση έγινε ήδη τον Ιανουάριο και τώρα συζητάμε για την πρώτη δημερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας. Η συμφωνία αυτή κανονικά θα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος θα είναι ο πολιτικός διάλογος, ο δεύτερος η συνεργασία και ο τομεακός διάλογος που περιλαμβάνει την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη συνεργασία και την ε, συνεργασία ε, σε εμπορικά θέματα. Φυσικά, αν μπήκαν σε λεπτομέρειες, ε, παρατηρεί ότι Αφενό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο ε, εξαγωγικό εταίρο τη Κούβα, είναι ο μεγαλύτερο ε, ξένο επενδυτή, αλλά τα ποσά είναι ακόμα χαμηλά. Δεύτερον, τα εμπορικά στοιχεία αυτού του πολιτικού ε, της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας είναι περιορισμένα τα εμπορικά και τα επενδυτικά στοιχεία. Πολλά ζητήματα αφορούν τη διευκόλυνση ε, των διοικητικών διαδικασιών, των τελών, αλλά των δασμών, αλλά ούτε η άλλη πλευρά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για την εκπόνηση κάποιου είδους συμφωνίας ελευθερών συναλλαγών, όπως συνήθως γίνεται ε, και σε άλλες χώρες της περιοχής. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν ε, μας δείχνει ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες συμφωνίες όπως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την Καρυβίκη. Ε, όταν βλέπει κανείς το μονοπόλιο ε, του εξωτερικού εμπορίου, ε, οι εισαγωγές που γίνονται με κρατικές άδειες, τα προβλήματα είναι πολύ απτά όσον αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου. Η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, παρότι παρατηρούνται κάποιε εξελίξει. Να επισημαίνω τι νέε δυνατότητε αυταπασχόλησης, για παράδειγμα, και θυμάμαι, το είπαμε την, περασμένη φορά, το 25% τη γη βρίσκεται στα χέρια των κουενταπροπίστε. Αυτό σημαίνει ότι παράγουν άνω του 50% των τροφίμων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και για τους άλλους τομείς. Πολλά λοιπόν, πολύ μεγάλο περιθώριο για εξέλιξη. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αλλάζουν, αλλά αργά μας λένε οι υπερογνώμονες. Αποτελεί στόχο της κυβέρνησης η προσέλκυση ε, περίπου 2,5 ε, δισεκατομμυρίων ε, άμεσων εξωτερικών επενδύσεων ετησίως ως κίνητρο ε, για να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη άνω του 5%. Έχουμε ήδη 250 κοινοπραξίες που υπάρχουν κυρίως από Ισπανία, Ιταλία, Καναδά και Βενεζουέλα. Από την άλλη όμως οι συνθήκες πλαίσιο για τις άμεσες ε, εξωτερικές επενδύσεις δεν είναι εύκολες. Ε, οι κανόνες για παράδειγμα απασχόλησης, ε, ο κρατικός έλεγχος των αδειών εισαγωγής και εξαγωγής δημιουργούν προβλήματα και έτσι βλέπουμε ότι ο αριθμός των επενδύσεων από το 2005 συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας της ειδικής ζώνης Μάρια ε, δεν έχουν ε, σημειώσει την εξέλιξη που θα θέλαμε να είχαμε δει. Από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός, η Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας αποτελεί μια αφετηρία για ανάπτυξη εμπορικών ε, και λοιπόν σχέσεων. Θα έχετε διαβάσει την γνωμοδότηση που, εκπονούσα, θα την έχουμε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα την προθεσμία υποβολή τροπολογιών και ήθελα απλά να επισημάνω όπως και στην προηγούμενη συζήτηση τον Ιανουάριο ότι καλωσορίζουμε αυτή τη νέα συμφωνία και ότι αναμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα σεβαστούν το ρόλο του Κοινοβουλίου και θα μας ενημερώνουν έγκαιρα καθώς επίσης και πριν από την υλοποίηση τέτοιων συμφωνιών ε, ότι θα δίνουν τη δυνατότητα στο κοινοβούλιο να δώσει το πράσινο φως. Στη γνωμοδότηση αυτή μιλάμε για το οικονομικό σύστημα, την ανάγκη ανάπτυξη του εμπορίου και την απελευθέρωση των άμεσων ξενεπενδύσεων, ε, την απελευθέρωση των εξαγωγών να αναφέρουμε και τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Πολλά ε, πρέπει να εξελιχθούν και καλωσορίζουμε και τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνεται σε μια από τις βασικές ε, τυπικές ρήτρες της συμφωνίας αυτής. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Απομένουν πολλά να γίνουν όπως τα δικαιώματα των ε, συνδικάτων, η προστασία του περιβάλλοντος, προσωπικά θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Πριν από μια μισή-δυο εβδομάδες έγινε μια ακρόαση με ένα πολιτικό ίδρυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εγώ ήμουν ο πρόεδρος και ένας από τους προσκεκλημένους, ε, η κυρία Μπάρτα Σολέα, η οποία έλαβε το βραβείο Ζαχάροφ το 2005, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει, δεν δηλαδή της το επέτρεψαν. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, οπότε πρέπει να επισημάνουμε ότι χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη ε, για τον πολιτικό αυτοδιάλογο και πρέπει να περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ο κ. Βαλέσσα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Κάποια στοιχεία εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Το σημείο 2 περιγράφει την πρακτική μη εφαρμογή των εμπορικών ή επενδυτικών διατάξεων πριν δώσει το πράσινο φως ε, ε, το Κοινοβούλιο θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί ή να επεκταθεί σε όλες τις διεθνείς μας ε, συμφωνίες. Με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στο σημείο 6 είναι σημαντικό Σίγουρα η Κούβα πρέπει να ε, σέβεται όλους τους κανονισμούς του Διεθνούς ε, Οργάνωση Εργασίας ώστε να αποφεύγει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό που είπατε εσείς τελευταίο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κοινοβούλιο μας απονέμει ετησίως το βραβείο Ζαχάροφ και όπως είπατε η κυρία Ζολαρή δεν, δεν μπορούσε να ταξιδέψει την περασμένη εβδομάδα. Οπότε είναι καθήκον μας να υποστηρίξουμε τη μάχη για την ελευθερία, να διασφαλίσουμε ότι οι καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα ε, θα ε, αποδοκιμάζονται διότι οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τεράστιο τίμημα παρενοχλούνται οι οικογένειές τους φυλακίζονται ε, κατεβαίνουν σε απεργίες πείνας άλλοι χάνουν τη ζωή τους υπό συνθήκες μυστήριες Οπότε τελικά πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Ποιος υποφελείται από αυτή τη συμφωνία και ελπίζω να μπορούμε να απαντήσουμε ο λαός της Κούβας εποφελείται όχι το καθεστώς. Αυτός είναι ο σκοπός, όχι το καθεστώς που τους καταπίεζε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεταφέρω τα σχόλια στον αδερφοντήτα. Μετά από 20 χρόνια της κοινή θέσης η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε νέα προσέγγιση απέναντι στην Κούβα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα συνεργασία, διάλογο και εμπορικέ σχέσεις. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για τα όσα αναφέρει σε σχέση με την βελτίωση της ζωής των Κουβανών κάτω από την περίοδο. Η Κούβα περνάει όμως όσο και αν εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τις αλλαγές αυτές, η Κούβα θα προχωρήσει μόνο αν σε αυτές συμπεριλαμβάνει όλους τους Κούβανους και αν ανοίξουν νέες ευκαιρίες ε, για την Κούβα. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Η συνεργασία, το άνοιγμα των αγορών μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαρατηθούμε από τις αξίες μας. Κάθε άλλο δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, συγγραφείς διώκονται. Και μάλιστα περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να στηρίξουμε μια συμφωνία μόνο αν αυτή βελτιώνει τη ζωή των κουβανών. Και για να γίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ελέγξει καλύτερα την ε, εφαρμογή των υποχρώσεων ε, που έχει αναλάβει η Κούβα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να γίνουν περισσότερα επίσης για την ελευθέρωση της οικονομίας κανόνες για την απασχόληση, ιδιωτικές εταιρείες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν δικαιώματα και αυτό εμποδίζει την Κούβα να προχωρήσει. Πρέπει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα με την υλοποίηση της νέας αυτής συμφωνίας. Θα υπάρξουν τροπολογίες για να ενισχυθεί το κείμενο, το οποίο όμως πηγαίνει πιστεύω προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Κουτιέρεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τις εξαιτίας των αλλαγών, των ε, ιστορικών ακριβώς αλλαγών που γίνονται στην Κούβα τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 2011 και μετά. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια εμπορική συμφωνία, αλλά με μια πολιτική συμφωνία και συμφωνία συνεργασίας με την Κούβα. Άρα θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έπαψε πια να ισχύει η κοινή θέση το 1996, θέλουμε να συνοδεύσουμε την Κούβα σε μια δημοκρατική διαδικασία με βαθιές αλλαγές στη χώρα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η πολιτική αυτή συμφωνία να τους αναφέρει τους στόχους αυτούς, ότι είναι πολιτική δηλαδή. Σε μια στιγμή που, όπως είπα, είναι ζωτική σημασίας. Πολλά μάτια από διάφορα σημεία του πλανήτη μας έχουν στρέψει την προσοχή τους πάνω στην Κούβα. Επίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε ε, ρητορικές έτσι συζητήσεις για το τι κάνουν 22 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα διμερός. Η συμφωνία αυτή, η πολιτική και η συμφωνία συνεργασίας, έχει την πρόθεση και να επηρεάσει θετικά τις αλλαγές, αλλά επιπλέον να προσφέρει και ένα πλαίσιο νομικής σταθερότητας, αντικειμενικότητας πέρα από τις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν, έτσι αλλιώ έχουν διπλασιαστεί από το 2009 μέχρι το 2015. Συνεπώς, προσπαθούμε με την έκθεση αυτή να σημειώσουμε ποια είναι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δεν πρέπει να ακολουθεί τα όσα κάνει το Συμβούλιο ή οι χώρες μέλη, πρέπει να έχουμε τη δικιά μας πολιτική τοποθέτηση υπέρ του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και να επωφεληθούμε από αυτήν την ιστορική σημασία στιγμή στις σχέσεις μας με την Κούβα. Πιστεύω επίσης, όπως είπα ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή αυτή, και θέλουμε να δούμε μετά τις αλλαγές στις Ηνωμένε Πολιτείες τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με την Κούβα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και από πλευράς ε, Ρωσίας ή Κίνας απέναντι στην Κούβα. Μην ξεχνάμε δηλαδή τον γενικότερο γεωπολιτικό χάρτη. Άρα λοιπόν η Κούβα πρέπει να είναι ισχυρή και αυτόνομη. Εμείς να επιμείνουμε στις αρχές μας και τις αξίες μας απέναντι στη διεθνή κοινότητα όπως πάντα κάναμε με όλες τις συμφωνίες που υπογράφουμε. Συνεπώς, ναι υπέρ της πλήρους δημοκρατίας, βελτίωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, βελτίωση επίσης της προστασίας των εργαζόμενων και των δικαιωμάτων τους, βάσει των συμφωνίων και των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ναι, υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεπώς, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται και το έχει ήδη δείξει αυτό η δικιά μου πολιτική ομάδα σε όλες τις συμφωνίες. Εμείς σαφώς και είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά στη συμφωνία αυτή πιστεύουμε ότι προσφέρει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Γι' αυτό δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται νέος χάρτης πορείας, όπως έχει γίνει σε άλλες συμφωνίες που είναι καθαρά εμπορικές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες. Συνεπώς, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την πορεία αυτή της Κούβας προς μια πιο κανονική κατάσταση και να χρησιμοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή ως εργαλείο για βελτίωση της κατάστασης στην κοινωνία. Νομίζω ότι είμαστε γενναιόδοροι, ισορροπημένοι, έξυπνοι, οπότε μπορούμε να μην κοιτάμε μόνο τις διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας, αλλά να μην ξεχνάμε γενικότερα την ιστορία μας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ιγνάσιο Ρανιέλ, παρακαλώ. Την κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν θα μακρηγορήσω, ήθελα απλά να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, η Κομισιόν συμμερίζεται την ανάλυση του εισηγητή όσον αφορά τις εμπορικές διατάξεις. Πράγματι δεν περιλαμβάνουν ε, πραγματική ουσία ουσιαστικά. Ε, η Κούβα παραμένει ε, στο πλαίσιο του πλέον ευνοημένου κράτους, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ωστόσο κάποια πράγματα περιλαμβάνουν ενδιαφέρον τη συμμετοχή της Κούβας στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Φυσικά αν από κουβανικής πλευράς υπάρξει βούληση να εφαρμοστούν τέτοιες ε, ε, διατάξεις. Τώρα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο έθεσαν ε, ουσιαστικά όλοι οι ομιλητές, να υπενθυμίσω ότι η PDCA προβλέπει διάλογο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, Υπάρχει μια συγκεκρι... ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο σκοπός της PDC είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα δώσει δυνατότητα ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβα ε, και βελτίωση της συνεργασίας τους. Αποτελεί ένα εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να βρεθεί σε καλύτερη θέση ώστε να συνοδεύσει τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Κούβα ε, και να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντά μας. Η υλοποίηση της συμφωνίας θα αποτελέσει την πλατφόρμα για επικοδομητικό διάλογο επί διαφόρων ζητημάτων όπως αυτά που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την πρόθεση της δημοκρατίας. Όλα θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής, πόσο ενεργά θα ε, υλοποιηθεί και από τον δραστήριο ρόλο ε, των θεσμών που δημιουργεί η συμφωνία κάποια προσθήκη από τον Κρίστον Φίσνερ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφο μου τα είπε όλα. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα μα βοηθήσει να αρχίσουμε κάποια γενική συνεργασία σε όλου του τομεί με την Κουβά. Η στάση μα προ την Κουβά δεν έχει αλλάξει. Η αηφόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι στόχοι μα όσον αφορά την Κουβά. Έχουμε το νέο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει ήδη ξεκινήσει είχαμε κάποια ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, αλλά αναμένουμε ακόμα ε, ε, θεσμική του πραγμάτωση. Παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην Κούβα και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Κάτι άλλο πολλά υποσχόμενο είναι επίσης το ότι η Κούβα έχει εκφράσει την επιθυμία της για προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα. Ε, ώστε να μπορέσει να διατεθεί ένα ευρωπαϊκό κονδύλιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. είναι η άνοιξη μιας νέα φάσης στη σχέση μα. Χρειαζόμαστε υπομονή και επιμονή. Αλλά ελπίζουμε ότι το εργαλείο αυτό θα μας επιτρέψει να συνοδεύσουμε την κουβά προς μια πιο σύγχρονη και ανοιχτή κοινωνία προ όφελο ε, του λαού τη Κούβα και των ευρωπαϊκών λαών φυσικά. Ευχαριστούμε. Για το ECR θέλατε να παρέμβετε. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα ήθελα να πω ότι Στηρίζουμε τα βασικά πολιτικά μηνύματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη γνωμοδότηση. Θα υποβάλουμε κάποιες μικρές τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο βασικούς τομείς. Ο ένας φυσικά είναι το εμπόριο και ο άλλος είναι το γεωπολιτικό πλαίσιο. Και οι δύο τομείς είναι αρκετά σημαντικοί το διεθνές εμπόριο αυτή τη στιγμή είναι σε περιορισμένο βαθμό, είναι περιορισμένη σημασία για την ε, κουβανική ε, οικονομία, αλλά πρέπει να εξεταστεί το θέμα της υπερβολικής γραφειοκρατίας, ε, της έλλειψης διαφάνειας και σίγουρα το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Επίσης, υπάρχει ευρεία διαφθορά και παράνομος οικονομικός τομέας ε, η σκιώδης οικονομία και όσον αφορά το γεωπολιτικό πλαίσιο όλοι γνωρίζουμε καλά τι συμβαίνει εκεί. Περιμένουμε πιθανές αλλαγές ε, στην ηγεσία της Κούβας. Και υπάρχει κρίση στην Βενεζουέλα που επί πολύ καιρό ήταν βασικός προμηθευτής της Αβάνα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Έτσι λοιπόν μπορεί να δούμε αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με την Κούβα. Επίσης, πιθανότατα να υπάρξει επανεξέταση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και να ακολουθηθεί κάπως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι κατά την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε το γενικότερο πλαίσιο. Όπως σας είπα και πριν, ε, όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε στις τροπολογίες μας ε, και προσλέπω στην επικοδομητική συνεργασία. Όπως πάντα, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος και παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας και επιτρέψτε μου μία παρατήρηση από συζητήσεις που είχα αλλού θα ήταν ωραίο, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, να έχουμε επαφές όχι μόνο με την κυβέρνηση, αλλά και να έχουμε επαφές και με την κοινωνία των πολιτών. Πρόεδρος, πράγματι νομίζω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Όπως ήδη υπόθηκε, η προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι τούτη η Παρασκευή, 5 Μαΐου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. και να σας θυμίσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά, διότι έχουμε πρόβλημα χρόνου. Παρασκευή 5 Μαΐου, τροπολογίες στα αγγλικά παρακαλώ. Και φτάνουμε στο σημείο 11, την επόμενη έκθεση του κυρίου Μπούγκε. Γενικός προϋπολογισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018. Παρακαλώ. Ε, δεν ε, προβλεπόταν η παρουσία του κυρίου Μούρεσαν ε, ως εισηγητή επί της ουσίας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έχουμε αρκετό χρόνο. Καταρχάς, προφανώς όλοι γνωρίζετε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου η διαδικασία μπλοκαρίστηκε από την Ιταλία και αυτή τη στιγμή μπλοκάρεται η ολοκλήρωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν αυτό θα λυθεί γρήγορα μετά τις εκλογές. Γι' αυτό επικρατεί αβεβαιότητα, διότι ε, το πακέτο αυτό, η δέσμη μέτρων, θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2018. Άσχετα από αυτό όμως είναι νομίζω απαραίτητο να ξαναεξετάσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές που υιοθετήσαμε στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά τη γνώμη μου το άρθρο 19 για την μεταναστευτική κρίση, το άρθρο 21 για την πολιτική γειτονία και τις συμφωνίες σύνδεσης, το 25 για χρηματοδότηση των ειδικών μέσων, και επιπλέον το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων, ε, όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Με βάση την προηγούμενη ε, έκθεση όπου μιλήσαμε για την ε, διαφθορά, ο συνάδελφος Σένφελ ανέφερε το θέμα αυτό. Θέλουμε σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών με το εμπόριο. Πώς θα το κάνουμε αυτό, βοήθεια προς τον προϋπολογισμό ή μήπως υπάρχουν προγράμματα πιο αποτελεσματικά από ότι η άμεση χρηματοδότηση. Διότι αλλιώς απλά σπαταλάμε χρήμα χωρίς να μπορούμε να το αιτιολογήσουμε κιόλας. Επίσης, ε, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το Brexit, ε, την ευελιξία στον προϋπολογισμό και ε, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στο άρθρο 26. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να συμπεριλάβουμε κάποια από τα θέματα αυτά. Και νομίζω επίσης ότι ε, η ανακοίνωση της Επιτρόπου Μάλμστρομ, ε, τώρα που έχει παγώσει η Συμφωνία του Ειρηνικού Ωκεανού από τον πρόεδρο Τραμπ, θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως θέλουμε εντατικοποίηση των εμπορικών ε, συζητήσεων ε, στον τομέα αυτών. Βρισκόμαστε λοιπόν σε προκαταρκτικό στάδιο, ακόμα δεν έχω καταγράψει τίποτα. Είμαι διατεθειμένος να ακούσω τις απόψεις των ε, συναδέρφων. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον Γενικό Εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κύριο Μουρεσάν και του δίνω κατευθείαν τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που με υποδέχεστε εδώ σήμερα. Ήρθα για να παρουσιάσω στους συναδέρφους τις κύριες προτεραιότητες για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για του χρόνο έτσι όπως εγκρίθηκαν από κοινού στην έκθεσή μου για τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου με μεγάλη πλειοψηφία στο Στρασβούργο. Αλλά πέρα από τις κύριες προτεραιότητες θέλω να ακούσω από τους συναδέρφους της Επιτροπής αυτής ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τις εξελίξεις επιτόπου για τα θέματα που είναι δικιά σας αρμοδιότητα και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πάντα στα θέματα που είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Υπάρχουν δύο κυρίω προτεραιότητες πάντως στον ε, προπολογισμό. Το ένα είναι η οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και το δεύτερο είναι η ασφάλεια των πολιτών. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες έτσι κι αλλιώ. Και γιατί πιστεύω ότι ακριβώς αυτό περιμένουν και από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δουλειά, έτσι, θέση εργασία και ασφάλεια. Πώ θα τα πετύχουμε. Απασχόληση πρώτα απ' όλα. Πιστεύουμε ότι είναι κυρίω ο ιδιωτικό τομέα, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που δημιουργούν θέσει απασχόληση. Άρα, προτεραιότητά μα είναι να του προσφέρουμε μια ισχυρή οικονομία, αξιόπιστη για του επενδυτέ. Άρα, υποδομέ, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη των νέων, όλα αυτά υπέρ της απασχόλησης. Horizon 2020, Connecting Europe Facility, διευκόλυνση για το δέοντα στην Ευρώπη δηλαδή, υποδομές, κόσμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και το πρόγραμμα έρασμο. γιατί δεν πρόκειται μόνο για ανταλλαγή φοιτητών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν από την έρευνα ότι πάνω από 60% των εργοδοτών εκτιμούν όλος ιδιαίτερος ε, τους υποψήφιους να πιάσουν δουλειά σε επιχειρήσεις τους αν αυτοί έχουν περάσει από μια τέτοιου είδους διεθνή εμπειρία. Άρα βοηθάει και το έρασμο στο να βρει κανείς δουλειά. Επίσης και στην αναθεώρηση των, των δημοσιονομικών προοπτικών υπήρχε το θέμα να προσθέσουμε 1,2 δισεκατομμύρια στο τωρινό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπέρ των νέων. Αν ε, διαβάσουμε την ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου βλέπουμε ότι χρειάζεται κάποια αναβάθμιση το πρόγραμμα αυτό, οπότε χρειάζεται και παραπάνω πρικοδότηση. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη προτεραιότητα που είναι η προστασία των πολιτών, η ασφάλεια. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση. Τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετά, γιατί ήδη από την αρχή της ε, εφτετούς περίοδου χρειάστηκε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα που μας έχουν μείνει λίγα. Οπότε ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα λίγα που μας έχουν μείνει. Οπότε το πρώτο είναι να ετοιμάσουμε προπαρασκευαστικές δράσεις για την άμυνα, κάτι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι μπορεί να βοηθήσει την έρευνα στην άμυνα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε 28 φορές χρήματα για το ίδιο πράγμα, για την ίδια έρευνα στις 28 χώρες μέλη. Καλύτερα μία φορά να τα συγκεντρώσουμε όλα και αυτό να γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Frontex, τη Europol, τη Eurojust, την EASO, που έχουν να κάνουν με θέματα ασφάλειας. Έτσι θα προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα και έτσι επίσης θα έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών όσον αφορά την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο όπλων, εμπόριο ανθρώπων, λαθροδιακίνηση κλπ. Και έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε καλύτερα και την γειτονιά μας, τις γειτονικές μας χώρες. Βλέπουμε να υπάρχει μια πιο επιθετική ρωσική ομοσπονδία τον τελευταίο καιρό, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως επίσης και για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πέρυσι το Μάιο είχαμε πάει στο Λίβανο και την Ιορδανία και είπαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της μετανάστευσης. Γιατί, γιατί φεύγει ο κόσμος από τις χώρες του, γιατί η υγεία, η εκπαίδευση, το νερό, οι υποδομές, η ασφάλεια δεν είναι καλά εκεί. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της μετανάστευσης και στις δικές μου κατευθυντήριες γραμμές το λέω και γιατί πρέπει να επενδύσουμε επίση σε αυτέ τι χώρε, γιατί μπορούμε περισσότερα να κερδίσουμε από ένα ευρώ εκεί παρά από ένα ευρώ υπέρ των ανθρώπων αυτών όταν αυτοί έχουν ήδη έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χίλια ευρώ το χρόνο ανά άτομο πρέπει να δώσουμε εκεί, ενώ αν είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερα στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία θέλουν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι γιατί λένε ότι άμα τελειώσει ο πόλεμος θα γυρίσουμε στις χώρες μας. Και αυτά για τους πρόσφυγες. Τώρα, κάτι άλλο. Αναθεώρηση του πλαισίου πολιτού, του πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου 2014 2020. Ε, Το 2013 πολλές ε, εξελίξεις που είχαμε τότε, τρομοκρατία, ασφάλεια, μετανάστευση, ε, ήταν προκλήσεις που δεν καταφέραμε να προλάβουμε. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία μέσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στο τίτλο 4 είχαμε 1,5 δισεκατομμύρια επιπλέον 270 εκατομμύρια για το εξωτερικό εύση, 200 εκατομμύρια επίσης για τη μακροοικονομική αρρωγή και βέβαια η επέκταση της δανειστικής εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προχωρήσαμε στο Κοινοβούλιο εμείς έγκαιρα. Τι έγινε στο Συμβούλιο όμως την προηγούμενη εβδομάδα που το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έπρεπε να τον κρίνει, το Ενωμένο Βασίλειο το έχει εμποδίσει το θέμα να προχωρήσει και αυτό θα το κάνει μέχρι τις Βρετανικές εκλογές τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο για μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Στον ε, τίτλο 4 αλλά και αλλού και για το κόσμο που είναι υπέρ των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων 200 εκατομμύρια παραπάνω είχαμε πει για το Horizon 2020 έρευνα ε, απασχόληση για τους νέους είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εγκριθούν όλα αυτά. Και τέλος για τα trust funds, τα κατεπιστεύματα. Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το θέμα, γιατί ναι, ήταν πήγον, έπρεπε να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα κάτω από δύσκολε συνθήσεις και δημιουργήθηκαν τέτοια trust funds, αλλά ως αρχές επί του προπολογισμού να μαθαίνουμε από τον τύπο ότι πήγαν τα 500 εκατομμύρια για την Τουρκία και να καταλάβουμε μετά ότι θα ήταν ένα δισεκατομμύριο, αυτό είναι απαράδεκτο. Έγινε μία φορά κάτω από έκτακτες συνθήκες, αλλά είναι σαφές ότι η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τα trust funds. Και τι είδαμε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κληθούν στα συμβούλια των trust funds προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό είναι θετικό. Παραμένει όμως Παραμένει ένα θέμα. Πρέπει να μπορούμε να προλάβουμε τα πράγματα πολύ περισσότερο από ό,τι το κάναμε το 2013 και να υπάρχει φρέσκο χρήμα για νέες προτεραιότητες οι χώρες 170 εκατομμύρια μόνο βάλανε ως περιθώριο. Για πολλά προγράμματα, ε, εκπαίδευση για παράδειγμα, χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα. Οι υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών επίση που στηρίζουν τον κόσμο επιτόπου πρέπει να ξέρουν ότι τα χρήματα τα οποία πολιτικά τους υποσχεθήκαμε θα τα πάρουν την επόμενη χρονιά. Αυτά από τη δικιά μου την πλευρά, Πρόεδρε. Κατά τα άλλα, η επίσκεψή μου εδώ θέλω να αποτελέσει το ξεκίνημα συνεργασίας μεταξύ μας. Τέλη Μαΐου θα έχουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εννοείται ότι θέλω να γνωρίζω την άποψη της Επιτροπής σας. Προσβλέπω επίσης τη γνωμοδότηση που θα ετοιμάσει η δικιά σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο Ράιμερ Μπέγκε, το έχει αναλάβει. Συμμετέχει και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Οπότε θα είμαστε σε επαφή όλη τη χρονιά. Και για τα πιλωτικά προγράμματα ξέρω ότι έχετε δύο. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα εξετάζουμε, τα έχουμε στείλει στην Κομισιόν για προαξιολόγηση. Αν υπάρξει ένα α ή ένα β από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θετική αξιολόγηση δηλαδή, θα κοιτάξουμε και εμείς να τα συμπεριλάβουμε. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας αυτή κύριε Μουρεσάν. Συνάδελφοι, μας τελειώνει ο χρόνος, μας πιέζει ο χρόνος. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομα. David Μάρτιν, παρακαλώ. Ε, πράγματι θα είμαι σύντομος. Ε, θα μιλήσω εκ μέρους ε, της ε, σκιώδους εισηγητριάς μας. Λέει λοιπόν ότι η εμπορική πολιτική είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα εργαλεία στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη σε τρίτες χώρες, να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και ο γενικός προϋπολογισμός του χρόνου θα πρέπει να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιδιώξει ε, φιλόδοξο εμπορικό θεματολόγιο. Τονίζουμε τη σημασία της σωστής εφαρμογής και ζητάμε κατανομή των απαραίτητων πόρων για την καλύτερη παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών γραμμή του προϋπολογισμού θα πρέπει να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην προσπάθεια τους για διεθνοποίηση. Εάν ε, δεν τα διασφαλίσουμε αυτά, τότε δεν θα αξίζει καθόλου όλη η δουλειά που έχουμε κάνει. Θα πρέπει λοιπόν ε, με προγράμματα να επιτρέψουμε αυτές τις επιπλέον δυνατότητες. Επίσης, ε, όσον αφορά τη μετανάστευση, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εμπορικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται και Επίσης θα ήθελα να αναφέρω το πρόγραμμα της Μακολάδα και την πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων. Για να έχουμε πραγματική αλλαγή χρειαζόμαστε όχι περισσότερα λόγια αλλά τα απαραίτητα μέτρα για να επιφέρουμε την αλλαγή. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι άλλο θα έχει γράψει αυτά. Δεν έχω συντάξει εγώ τα αγγλικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ θέλετε... Ε, κύριε Σαγρατήλ, όχι. Ε, Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα όσον αφορά το Ταμείο Μαντάτ και τα άλλα εργαλεία πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, θα έχουμε την δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτά στην σχετική ομάδα εργασία. Σε σύντομα όμω για το εμπόριο, διότι εδώ επικεντρωνόμαστε σήμερα, βλέπουμε ότι ε, όχι μόνο έχουμε πιο φιλόδοξη προσέγγιση την οποία επικροτούμε, αλλά ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά τις γεωπολιτικές σχέσεις, ε, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει ως ευκαιρία και να τις εκμεταλλευτεί. Στο παρελθόν έχω ζητήσει επανειλημμένα και δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έχω ρωτήσει λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επαρκή σπόρους, δυναμικό, ε, ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και αρκετό προϋπολογισμό διότι όχι μόνο έχουμε αύξηση στον όγκο των διαπραγματεύσεων, υπάρχει επίσης σημαντική αύξηση στον έλεγχο από το κοινό, ε, απέτηση για περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή. Οι ικανότητες ενός διαπραγματευτή μπορεί να είναι καλές για τις διαπραγματεύσεις, αλλά μπορεί να μην ε, αρκούν ή να μην είναι κατάλληλες για τις επαφές με τους ενδιαφερομένους. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το δυναμικό σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά την συμμετοχή, την ε, ε, διάδοση των πληροφοριών κλπ. Ρωτώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλά εξοπλισμένη. Επίσης νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν διότι εκεί να δίνουν εντολή στην Επιτροπή να τα κάνει όλα αυτά στο όνομα όλων μας, διότι νομίζω ότι αυτό μας κάνει πιο ισχυρούς σε έναν κόσμο που αλλάζει. Θα πρέπει επίσης οι κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη να εξηγήσουν στους πολίτες τους, στους ενδιαφερομένους κύκλους, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να φροντίσουμε να χρηματοδοτούνται οι δράσεις που ζητώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μου μήνυμα και τέτοιου τύπου τροπολογίες να περιμένετε από την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Χέλμουτ Παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση, την εισαγωγή σας, που ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή εισαγωγή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές. Καταρχάς, έχουμε το Brexit και όλα τα σχετικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον όλες ε, τις δραστηριότητες που περιγράφουμε και στον τομέα του εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν μάλλον να οδηγηθούμε σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι τμήμα του προϋπολογισμού θα προέρχεται από αυτούς τους ίδιους πόρους. Κάτι που με οδηγεί στη δεύτερη μου παρατήρηση. Η ομάδα μου μάλλον δεν συμφωνεί να μεταφέρουμε υπερβολικά πολλά θέματα στον τομέα της ασφάλειας, ε, λέγοντας ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, την Frontex κλπ. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις ε, αιτίες της μετανάστευσης και το να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην νότιο-ανατολική γειτονία είναι πολύ κοντόφθαλμο. Ακούσαμε τα στοιχεία για την Κάνα οι εταίροι μας είπαν ότι πρέπει να επανεξετάσουν τη δυνατότητά τους να επικεντρωθούν στην διμερή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι ίδιοι άνθρωποι επιλέγουν ή τον Βορρά ή τον Νότο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ενισχύσουμε και τη δική μας ικανότητα να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και συμφωνώ με την Μαρίτα Σάκε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε όλα που διαπραγματευόμαστε να είναι καλά στηριγμένα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και με τον εισηγητή και να δούμε πώς η Εμπορική Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρατηρήσα του τους Πρασίνους όχι. Ωραία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Yes. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Θα, θα είμαι σύντομη. Στην παρούσα φάση, όπως γνωρίζετε, η πρόταση της Κομισιόν για τον προπολογισμό δεν έχει εγκριθεί ακόμη, οπότε μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου στο πλαίσιο της άσκησης ε, εκπόνησης πρότασης του προπολογισμού σε επίπεδο επιτροπής. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ήδη ότι πολλά από τα ζητήματα που αναφέρατε στη συζήτηση βρίσκονται ήδη μεταξύ, ήδη μεταξύ των προτεραιοτήτων που θα εξετάσουμε εμείς με τον πολύ μικρό μας ε, επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Πράγματι, η εμπορική ατζέντα επεκτείνεται διαρκώς. Αυτό αποτελεί πρόκληση για μας τόσο σε θέματα ανθρωπινών πόρων όσο και από δημοσιονομική άποψη. Έχουμε χαμηλό προϋπολογισμό λειτουργικό, αλλά χρησιμοποιούμε και άλλα εργαλεία σε περιφερειακό και δημερές επίπεδο τα οποία εξετάζουν την υλοποίηση και τη διαπραγμάτευση των εμπορικών μας ε, συμφωνιών. Εστιαζόμαστε στην παρακολούθηση επίσης των εμπορικών ε, συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε και ήδη φέτος Εάν ο προπολογισμό ε, εγκριθεί σύμφωνα με τα όσα έχουμε προτείνει, φέτος θα εστιαστούμε στην επικοινωνία και τις σχετικές δραστηριότητες, ε, ειδικότερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε συμφωνήσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, θα πρέπει να είναι το κύριο σημείο εστίαση των δραστηριοτήτων επικοινωνία μα, διότι αυτέ θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο τι συμφωνίε που εμεί δεν πραγματευόμαστε. Επίση, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία στι δραστηριότητε αξιολόγηση τόσο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όσο και αφού υλοποιηθούν οι συμφωνίες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υλοποιούνται σωστά, αλλά και για να ανεχνεύουμε πιθανές ανάγκες περαιτέρω εξέλιξης ή ανάπτυξης σε συμφωνιών που ήδη ισχύουν. Επίσης, Μαζί με άλλες γενικές διευθύνσεις θα εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη διεθνή τους διάσταση τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Σημαντικό τομέας για μας ε, ε, το λαμβάνουμε υπόψη στις συμφωνίες μας αλλά και σε διάφορα εργαλεία όπως το κόσμο που ανέφερε ο εισηγητής της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Κύριε Μπέγκε, θα θέλατε να σχολιάσετε. Όχι, Μάλλον όχι τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ε, δύο παρατηρήσεις. Ο συνάδελφο ε, Σόλτ έχει δίκιο. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι σύστημα ιδίων πόρων θέλουμε. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συζητηθεί για τις επόμενες, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα πιο διαφανές. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων για τον Brexit να δούμε και τι αποζημίωση θα δοθεί. Και θα έχουμε να κάνουμε πολλούς πολύπλοκους υπολογισμούς. Θα πρέπει λοιπόν εγκαίρως να θέσουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και συμφωνώ με την συνάδελφο Σάκε. συζητήσαμε τις ε, εξελίξεις ε, στο πλαίσιο της Συμφωνίας ε, του Ειρηνικού. Αλλά θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει και τι δυναμικό έχει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τι θα χρειαστεί στις διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς και τελικά ε, ποια θέματα θα θεωρηθεί ότι έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα. Θέλουμε σταθεροποίηση στις γειτονικέ μας χώρες ε, και οι εμπορικές συμφωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό διότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην παραμεληθούν κάποια θέματα λόγω κάποιων άλλων αναγκών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα είναι πολύ δύσκολες οι συζητήσει για τον προϋπολογισμό. Ε, άλλωστε έχουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τίθεται το ερώτημα θα ε, ισχύσει μέχρι το 2020 ή ε, θα ε, περιοριστεί χρονικά λόγω του Brexit. Ε, θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Την επόμενη φορά νομίζω θα το συζητήσουμε αυτό 19 ή 20 Ιουνίου. Ευχαριστώ τον Γενικό Εισηγητή που ήταν παρόν. Και μας εύχομαι καλή επιτυχία στις ε, περαιτέρω συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο σημείο 12. 25 λεπτά μας μένουν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να παρουσιάσουν ε, σύντομα τα επιχείρηματά τους. Το θέμα μας είναι η αναδιατύπωση του κανονισμού διπλής χρήσης και έχουμε την σχετική έκθεση και χωρίς πολλά πολλά δίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το σχέδιο ε, έκθεσης περιλαμβάνει 57 ε, τροπολογίες. Μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνονται πολλές, ε, αλλά σε μεγάλο βαθμό ε, επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένη τροποποίηση διατύπωσης που επανεμφανίζεται στο κείμενο. Σε τέσσερις ομάδες μπορούμε να χωρίσουμε τις τροπολογίες μας. Καταρχάς θέλουμε απλοποίηση για τους εξαγωγείς. Με αυτό σχετίζεται η, παράταση, η πρότασή μου για παράταση των ε, αδειών εξαγωγής. Και να αφαιρεθούν ε, κάποια, κάποιοι τομείς όπως ε, είναι η κρυπτογραφία ή τα εγκληματολογικά βοηθήματα. Επίσης, η ασφάλεια είναι ο βασικός πυρήνας αυτού του, κανονισμού και προτείνω φορτία χαμηλής, ποιο... Ε, χαμηλής αξίας ε, και μεγάλα προγράμματα να ε, αφαιρεθούν από τον κατάλογο. Όριο για την χαμηλή αξία είναι τα 5.000 ευρώ τον ε, μήνα, δηλαδή 60.000 ε, ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν είναι κάτι που σχετίζεται με την ασφάλεια και ε, τα μεγάλα έργα περιλαμβάνουν τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι κάτι που αφορά άμεσα την ασφάλεια μας. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικό για να γνωρίζει ότι εάν κάποιος έχει πυρηνικό εργοστάσιο δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσει και ε, πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά με την εξαγωγή ε, πυρηνικών αντιδραστήρων έχουμε ήδη κάνει το πρώτο βήμα. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι είναι λάθος να διευκολύνουμε την εξαγωγή αυτών. Επίσης, προτείνω να ελέγχεται ο τελικός χρήστης σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό αντίστροφα σημαίνει ότι ε, οι μεμονωμένες ε, άδειες ε, οδηγούν σε μεγαλύτερη υποψία και δεν είναι έτσι δυνατό να υπάρχει εγγύηση για τον τελικό χρήστη. Αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι. Η τρίτη ομάδα προτάσεών μου έχει να κάνει με την προβλεψιμότητα για τους εξαγωγείς μας. Αυτό μας το ζήτησε ο οικονομικός τομέας. Γι' αυτό θέλουμε πιο σωστούς, πιο ακριβείς ορισμούς για κάποιους βασικούς όρους όπως είναι η ιδέουσα επιμέλεια, το due diligence. Και όσον αφορά τον ορισμό των αγαθών που έχουν να κάνουν με την κυβερνοεπιτήρηση για να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια προγραμματισμού, θα πρέπει να εξετάζουμε ε, τα κριτήρια για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποια χώρα, πώς ε, και από ποιον εξετάζονται. Επίσης, κυβερνοεπιτήρηση ε, πλέον συμπεριλαμβάνεται στο νέο τομέα 1β του παραρτήματος. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί η απόρριψη των σχετικών αιτήσεων. Και στο πλαίσιο κάποιων διεθνών φόρουμ όπως είναι ο ΩΣΑ πόσο μπορούμε να έχουμε νέα διεθνή πρότυπα. Έχουμε μια σειρά κρατών μελών που ελέγχουν κάποιες τεχνολογίες επιτήρησης. Με τον κανονισμό αυτόν μπορούμε να έχουμε πιο συντονισμένη προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να δράξουμε την ευκαιρία αυτή. Αυτό βοηθάει και την ασφάλεια προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, στον κανονισμό αυτό υπερσπιζόμαστε τα συμφέροντά μας ε, στο εμπόριο και στην ασφάλεια. Με το σχέδιο αυτό προτείνω κάποιες διευκολύνσεις για τους εξαγωγείς ε, αλλά και κάποια ζητήματα που δυσκολεύουν. Ε, θέλουμε όμως να υπάρχει ασφάλεια προγραμματισμού, κάτι που είναι προς όφελος των εξαγωγέων. Πιστεύω ότι έχω βρει καλή ισορροπία. Ελπίζω να μπορέσετε να στηρίξετε την έκθεσή μου. Επίσης, σε λίγα λόγια για τις δικές μου τροπολογίες. Θα προτείνω κάποιες τροποποιήσεις στα παραρτήματα. Πιο σημαντική διάσταση εδώ είναι η διαγραφή της κρυπτογραφικής τεχνολογίας από τα παραρτήματα. Αυτό είναι πολύπλοκο διότι θίγονται διάφορα άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό χρειάζομαι σχετική εμπειρογνωσία προτού να μπορέσω να το κάνω αυτό στην πράξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκπροσώπους του οικονομικού τομέα με τους οποίους συναντήθηκα στο πλαίσιο της εκπόνησης ε, του σχεδίου ε, έκθεσης. Ε, στην ιστοσελίδα μου, καθώς ε, και επίσημα στην ε, ιστοσελίδα της, του Κοινοβουλίου μπορείτε να βρείτε τις επαφές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Λόγω της πίεσης του χρόνου, δύο λεπτά για την κάθε παρέμβαση. Παρακαλώ. Ο κύριος, ο κύριος Γασπάρη, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις παρατηρήσεις του Κρίστοφερ Φιέλνερ που είναι σκιώδης εισηγητής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση αυτή. Αγγίζει διάφορα ζητήματα, την ανάγκη αδιαφάνεια για όλου του ενδιαφερομένου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ελέγχου των εξαγωγών και των επιχειρήσεων. Ε, το ΕΛΚ ζητά ε, συνεκτικούς ε, και αναλογικούς ε, τελωνιακού έλεγχους των εξαγωγών ε, με διαφάνεια για τις ε, επιχείρησεις της Ευρώπης. Ωστόσο ανησυχούμε όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής και μας ανησυχούν ορισμένα από τα επτά σημεία που επισημαίνει ο εισηγητής. Η ρήτρα στόχου είναι ευρύτερη από την πρόταση της Κομισιόν η ρήτρα catch all, αν πρόκειται να υπάρχει τέτοια ρήτρα θα πρέπει να είναι ακριβής και να βασίζεται ε, ε, στην πρόληψη των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε παγκόσμιες ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Πρέπει να ε, έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα πολυμερή καθεστώτα. Μ' αρέσουν οι προτάσει του εισηγητή για επέκταση της, του χρόνου άδεια στα δύο χρόνια. Με ευχαριστή θα συζητήσω με τους ε, συνεισηγητές, ε, με τους κύριους συζητητές, όταν θα έχουμε περαιτέρω ε, προτάσεις. Τώρα, ο σκιώδης συζητητής των σοσιαλιστών πρέπει να πω ότι πρώτα απ' όλα, πρώτα η εκθέση του κύριου Μπούχνερ είναι θετική. Εμεί θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες η ρήτρα όλοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ενισχυθεί. Συμφωνούμε δηλαδή επί του θέματος αυτού. Δεν αρκεί να κάνουμε έκκληση για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να κάνουμε και πρακτικές συστάσεις για το πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα λεπτομερές εγχειρίδιο όπως έχουμε και για άλλες ε, περιπτώσεις. Ε, ε, θα υπάρξουν εμπειρογνώμονες που θα μας βοηθήσουν, οπότε θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την αξιολόγηση. Ε, όλα αυτά στο πλαίσιο του άρθρου 14. Όσον αφορά τη γενική ρήτρα για την τρομοκρατία, το πρόβλημα εκεί δεν είναι καθόλου το ίδιο. Το ότι ορισμένοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, από τους τρομοκράτες δεν είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Ε, επίσης υπάρχουν ήδη διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις υποθέσεις ανθρώπων που σχετίζονται με τρομοκρατικές οργανώσεις. και να ασκήσουμε τη δεωσα επιμέλεια. Επιθυμούμε επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλύτερη διαφάνεια, ό,τι δεν είναι εμπορικό απόρριτο. Μάλλον όσον αφορά τον ορισμό του εμπορικού απορρίτου και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Θα θέλαμε μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία και πιο αποτελεσματική και σε περισσότερα θέματα. Και επίσης και εκεί θα πρέπει να ελαφρύνουμε λίγο το φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις και εκεί μπορούμε να επιδείξουμε κάποια καινοτομία. Αυτά. Ο κύριε Ζαχράντιλ ε, για το ECR. Εκ μέρου του συγητή μα ε, που δεν μπορεί να είναι εδώ τώρα. Θέλω να πω ότι γενικώ το σχέδιο αυτοέκθεσης είναι αποδεκτό. Έχουμε διευκρινήσει στις τροπολογίες, αλλά δεν στηρίζουμε την πρόταση του συγητή για διαγραφή της ε, άδεια του τελευταίου σχεδίου, γιατί πιστεύουμε εμεί ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο γενικό από την εξαγωγή νέων σχεδίων, έτσι όπως το βλέπει στενά ο εισηγητής. Και άλλα θέματα χρειάζονται διευκρίνηση, γιατί είναι αρκετά δύναμη διατύπωση για το ποιε είναι οι υποχρεώσεις των εξαγωγών που δεν διατυπώνεται πολύ ξεκάθαρα κάποια από αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι επιπλέον άχθος για αυτούς που ελέγχουν τις εξαγωγές ε, στα τελωνία για το κατσόλ, για παράδειγμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για διπλής χρήσης προϊόντα. Και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες από την ΑΦΕΤ και η γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ μπορεί να είναι χρήσιμα πράγματα έτσι ώστε ο κανονισμός να γίνεται κατανοητός πιο ομοιόμορφα και να προσφέρει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, κυρίως για τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία ελέγχου στο κυβερνοχώρο και το άρθρο 4 παράγραφος 1 για τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πάντως, ο κ. Λούνης και ο εισηγητής προσβλέπει σε συνεργασία με τον εισηγητή για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε και κυρία Σχάκη από το Άλντε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα είμαι σύντομη παρόλο που πολλά θα μπορούσε να πει κανεί εδώ. Γνωρίζουμε ότι η ενημέρωση του κανονισμού αυτού για τα προϊόντα διπλής χρήση είναι κάτι αναγκαίο για να λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές, ...στην πραγματικότητα στον κόσμο σήμερα, αλλά και νέου κινδύνου που εμφανίζονται. Κυρίω όμως έχουμε την επανάσταση στον τομέα της πληροφορικής και είναι αυτό το οποίο μας κάνει να θέλουμε την ενημέρωση αυτή. Επίσης τεχνολογίες εποπτείες γίνονται πιο μικρές, πιο φτηνές Άρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει στην Ευρώπη για το πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα, τέτοια τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που θα πρέπει να θέσει υψηλότερες προδιαγραφές στις εμπορικές της σχέσεις. Η τεχνολογία προχωράει κάθε μέρα και έχουμε δει ότι το σύστημα ελέγχου εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να εμποδίσει κάποιες από αυτές τις εξαγωγές ε, τεχνολογίας ώστε να φτάσουν σε χώρες όπου θα χρησιμοποιηθούν τελικά σε βάρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει υπόψη στο θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Χρειάζεται νομική ασφάλεια και βεβαιότητα αν θέλουμε ο κανονισμός αυτός να έχει τον αντίκτυπο που θέλουμε και να δεσμεύσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ε, πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση και εφαρμογή. Στην ΑΦΕΤ πρότεινα να διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο τον, ε, το θέμα του ελέγχου με τον κατάλογο των ε, μη περιλαμβανόμενων προϊόντων διπλής χρήσης πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Αλλά εδώ δεν αναφερόμαστε γενικά σε ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε σοβαρές παραβιάσεις, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασανισμοί κλπ. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή να διευκρινίσουμε τους ορισμούς που δεν έχει διατυπώσει ξεκάθαρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα η διευκρίνηση είναι το ένα βασικό. Το άλλο είναι να δούμε οι εθνικές αρχές τι κάνουν. Πολύ συχνά έχουμε δει ότι γίνονται ε, παράνομες ή τέλος πάντων αμφιβόλουν νομιμότητα σε εξαγωγές από τις χώρες μέλη. Τεχνικά μπορεί να μην ήταν κάτι παράνομο όταν έγιναν, αλλά ακριβώ γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αξιόπιστη και να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και να μην υπάρχει η αρχή σε θελοντική βάση μόνο ανταλλαγής πληροφοριών που θεωρούνται σημαντικές για τον άλλον. Πρέπει βέβαια να επιδείξουμε και ευαισθησία για πληροφορίες που προφανώς και δεν μπορούμε να μοιραστούμε πάντα με τους υπόλοιπους. Χρειάζεται πάντως ομοιόμορφη ερμηνεία και ισότιμη αντιμετώπιση. Να μην ρυθμίσουμε υπερβολικά επίσης, να μην έχουμε ελέγχου εκεί όπου δεν χρειάζεται. Είναι σημαντικό αυτό στα πλαίσια της έρευνας για την ασφάλεια και των δοκιμών. Και ο έλεγχος της αποκρυπτογράφησης είναι επίσης κάτι σημαντικό τον 21ο ε, αιώνα. Δεν μας κάνει πιο ευάλωτου, μας κάνει πιο δυνατούς. Τέλος, ευχαριστώ και τον εισηγητή και την Επιτροπή που υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται σαφήνεια και νομική βεβαιότητα. Ελπίζω επίσης το Συμβούλιο να επιδείξει συνεργασία για το θέμα αυτό και να υπάρξει ενημέρωση αυτή του κανονισμού όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε. Έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο στην εισηγήτρια από την ΑΦΕΤ. Μαρίν Μιρέ τώρα από την ε, ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι βάζουν τα ακουστικά τους βλέπω. Λέει στο Ολλανδικά η ομιλήτρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και συμφωνούμε και εμείς με αυτό. Έχουμε και θα ετοιμάσουμε και άλλες τροπολογίες. Χρειάζεται καλύτερη αναφορά όσον αφορά αυτήν την διπλή χρήση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Η πρόταση του εισηγητή να υπάρξει κατάλογος ε, τέτοιων ε, προϊόντων. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ομοιόμορφη μορφή. Και αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Επίσης να διευρυνθεί ο κατάλογος και να γίνει αυτό γρήγορα με προϊόντα το οποία ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται και είναι διπλής ε, χρήσης για διάφορα φίλτρα που χρησιμοποιούν στις τεχνολογίες, μπορούμε να δούμε τη νύχτα, Τέλος, θέλω επίσης εξάντε να γίνονται όλα αυτά και όχι ex post. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε ένα προϊόν, ένας μηχανισμός που θεωρούμε ότι είναι αμφιβόλου νομιότητας να μην επιτρέπουμε να υπάρχει εξαγωγή του. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τίτσιανα Μπεγκίν για το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συναδελφοί. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας ε, ε, εποπτείας. Μπορούμε να κατασκοπεύσουμε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να ελέγχουμε τηλέφωνα, να διαβάζουμε email και να επαληθεύουμε και τις μετακινήσεις ε, μέσω εφαρμογών στα smartphone. Αυτό που είναι σκανδαλώδες είναι ότι πουλάμε τέτοια μέσα σε δικτατορίες που έτσι συλλαμβάνουν και σκοτώνουν πολίτες τους. Η Ευρώπη πουλά τεχνολογίες επιτήρησης ε, προς παραβίαση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για παράνομες εξαγωγές, αλλά πολύ συχνά κάποιες επιχειρήσεις ε, απλά εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος, τα οποία πρέπει να κλείσουμε για αυτό το σκοπό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία ώστε να βοηθήσουμε τις τίμιες επιχειρήσεις που εξάγουν νόμιμα τα προϊόντα τους προς ε, δημοκρατικές χώρες. Ε, και να τι απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό βλέπω θετικά τι αλλαγέ του εισηγητή και τον συγχαίρω. Αφού οι περισσότερε τροπολογίε του με βρίσκουν σύμφωνοι. Σύμφωνο επίσης ε, την υπογράμμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το αίτημα προς τους εξαγωγείς ε, να μαθαίνουμε αν ό,τι εξάγουν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέκταση του κανονισμού για όλους τους τύπους εργαλείων, όχι μόνο των κινητών συσκευών, και διότι πολύ γενικά πολλές φορές ε, μιλάμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες. με κατά της εξαγωγής ε, τέτοιων προϊόντων σε παράνομα, ε, σε παράνομα κατακτηθέντα εδάφη και επίσης μ' αρέσει που έχουμε τον ορισμό για τις τρομοκρατικές ομάδες και συμφωνώ με την επέκταση της άδειας στα δύο χρόνια. Αυτό θα βοηθήσει από άποψη γραφειοκρατίας στις τίμιες επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι, πριν καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε μια εμπορική πολιτική που θα βασίζεται σε αξίες. Εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν εξάγει μόνο τεχνολογίες εχμής και ε, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει γενικά με την εμπορική πολιτική μας που να βασίζεται σε αξίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ, ποιος θα θέλει να πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανείς. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Χαιρόμαστε με την αποφασιστικότητα που δείχνει για ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπεύθυνο ε, να ε, παρεμποδίσει εξαγωγές ε, που οδηγούν ε, που υπονομεύουν την ασφάλεια και οδηγούν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίων. Συμμεριζόμαστε την ανάλυση ε, και τις απαραίτητες αλλαγές για την πολιτική ασφαλείας και θέλουμε να προσαρμόσει τα εργαλεία της Ευρωπαϊκή Ένωση όπως χρειάζεται και καθώς και τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών. Μας συγκινεί η μεγάλη υποστήριξη ε, της διάστασης της ανθρώπινης ασφάλειας που προτείναμε εμείς και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ε, ευρύτε, τα σημεία που αναφέρουν την ε, ε, παρακολούθηση ανθρώπων είναι θέματα ασφάλειας σημαντικά. Σημειώνουμε επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη νομική σαφήνεια Περιλαμβάνεται αυτό και στο σχέδιο γνωμοδότησης της ΑΦΕΤ και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία για να γίνει πιο σαφής η πρόταση όπου απαιτείται. Ειδικότερα, επανειλημμένως μετά από την υιοθέτηση της πρότασης έχουμε αναφέρει ότι είμαστε έτοιμοι για την εκπόνηση κατηδύρων γραμμών για τη διάσταση αυτή της ασφάλειας των ανθρώπων. Παρατηρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης διευρύνει την προσέγγιση για την ασφάλεια των ανθρώπων πέραν των ε, εμπόλεμων καταστάσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε μια στοχευμένη προσέγγιση ώστε να αποφευχθούν, ε, ε, αποφευχθεί εργασία εργασίας και στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι οι κρυπτογραφικοί έλεγχοι αν μη τι άλλο θα πρέπει να διευκολύνονται. Κάτι που αναφέρεται ουσιαστικά στην πρότασή μας σε κάποιο βαθμό. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι η έλεγχη η ασφάλειας των ανθρώπων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν ε, την ε, έρευνα στο διαδίκτυο. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία είμαστε διατεθειμένοι να μελετήσουμε περισσότερο. Τέλος, σημειώνουμε την έκκληση για μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνεια. Η πρότασή μας ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και με μεγάλη μας χαρά θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα συμβέσμο, έναν τρόπο για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα προωθεί τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα όπως αναφέρεται στην έκκληση του Κοινοβουλίου. Τέλος, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την ΙΝΤΑ, με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη προς ένα ε, πλαίσιο εξαγωγών ε, ανθεκτικό στο μέλλον. Αυτή την πρόταση ε, θα υποστηρίξουμε και εμείς στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπούχνερ. Θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένου της πίεσης χρόνου δεν θα απαντήσω σε κάθε παρατήρηση που έγινε, θα το κάνω όμως αργότερα. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε κιόλα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Μαΐου το μεσημέρι στις 12. Και στις 30 Μαΐου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα προβλέψουμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε εις βάθος. Στις 19 Ιουνίου θα, ψηφίσουμε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Κλείνω λοιπόν το θέμα αυτό. Ένα λεπτό διάλειμμα για να προχωρήσουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών.